Je vous propose que nous commencions. Donc le premier sujet à l'ordre du jour euh, est le... Καλημέρα. Ξεκινάμε με την έκθεση σχετικά με την ε, ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ριβελίνη για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Κύριε Ριβελίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι η καθήλια αρμόδια επιτροπή, να συμπεριλάβει στο σχέδιο ψηφίσματος που θα υιοθετήσει το Μάρτιο κάποια, κάποιες προτάσεις, τις οποίες έχω περιορίσει στο, που, που έχουν σαν στόχο να περιορίσουν στο ελάχιστο τις ε, συνέπειες ε, και τις παρενέργειες στην υγεία ε, των, της που εκπέμπουν οι σαρωτές σώματος, έστω και αν η ακνοβολία αυτή είναι ελάχιστη η πιο κατάλληλη, πλέον κατάλληλη λύση για την υγεία είναι η τεχνολογία που βασίζεται σε συστήματα επεξεργασίας εικόνας ανενεργών χιλιοστομετρικών κυμάτων που δεν εκπέμπουν καμία ακτινοβολία. Διότι από τις μελέτες που έχω διαβάσει βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για την υγεία. Δεύτερον, προτείνουμε σαν πιο κατάλληλη όμως λύση, σαν δηλαδή συμβιβαστική λύση αν θέλετε, μια πιο ισορροπημένη λύση, την ε, ε, λύση που βασίζεται σε συστήματα επεξεργασίας εικόνας ενεργών, ενεργών χιλιοστομετρικών κυμάτων αυτή τη φορά, που χρησιμοποιούν την μη ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία γενικά θεωρείται αυλαβής εάν η έκθεση όμως δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που ορίζονται στη σημερινή νομοθεσία. Τρίτον σημείο. Επισημαίνουμε ότι η τεχνολογία που βασίζεται στην οπισθοδιάχυση των ακτινών χ, εκπέμπει μια χαμηλή δόση ακτίνων χ. Γνωρίζουμε προφανώς ότι οποιαδήποτε έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία έστω και αν αυτή είναι χαμηλή ισχύω, μπορεί να έχει επιπτώσεις μακροπρόθεσμα στην υγεία λόγω του σορευτικού αποτελέσματος των ακνοβολιών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προτείνει να αποφεύγεται η χρήση αυτής, αυτής της τεχνολογίας, συγγνώμη, εξού και θα πρέπει οι ε, εκπομπές, η, η, ε, η έκθεση των, ε, εργαζομένων ή των ταξιδιωτών, των επιβατών, θα πρέπει να είναι όσο το πιο χαμηλές. Τέταρτον, υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία που βασίζεται σε ακτινογραφίε εκπέμπει υψηλή δόση ακτινών Χ και επομένω δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για, για το συστηματικό έλεγχο στο πλαίσιο τη εναέρεια ασφάλεια. Πέντε, ζητάμε όσον αφορά την χρήση σαρωτών σώματο με ακτίνες Χ, που είναι το σημείο 3, να χρησιμοποιούνται ειδικέ μέθοδοι, κυρίως για τους επιβάτες που είναι ευαίσθητοι στην ιονίζουσα εκνοβολία, όπως οι έγκυες ή τα παιδιά. Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις για τα άτομα με εμφυτευμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως οι βηματοδότες και οι απεινιδωτές. Και σημείο 6, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν σε τακτική βάση τις επιπτώσεις της έκθεσης, της μακροπρόθεσμης έκθεσης του σωρωτέ σώματος, να λαμβάνουν υπόψη τις νέες τεχνολογίες, τις νέες εξελίξεις συγγνώμη, και τις νέες τεχνολογίες και να ελέγχουν την ορθή εγκατάσταση, την ορθή χρήση και την ομαλή λειτουργία αυτών των συσκευών. Το σημείο 7 ζητούν από τα κράτη-μέλη να ε, προσφέρουν ε, στους επιβάτες σαφείς πληροφορίες και πλήρες πληροφορίες στα αεροδρόμια πριν ε, ξεκινήσει το ταξίδι, να τους ενημερώνουν δηλαδή για όλες τις πτυχές της χρήσης των σαρωτών. Γι' αυτό το τελευταίο σημείο, το σημείο 7, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο γνωμοδότησης, επειδή δεν, ήταν, δεν πρέπει να είναι ήταν μεγάλο το, το κείμενο, θα σας το προσθέσουμε και θα σας το δώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Φώστερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με όσα είπε ο κύριος Ριβελίνη. Και για να δούμε τα πράγματα στο πραγματικό τους πλαίσιο, αρχικά ήμουν εγώ η συγγήτρια ε, για το 23-20 μετά τις επιθέσεις της 11 ε, Σεπτεμβρίου. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και είναι μια δύσκολη. Εγώ είμαι πλήρες μέλος στην Επιτροπή Μεταφορών και πρέπει να ξέρετε ότι εκεί συζητιούνται διαφορετικά θέματα όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Εντελώς διαφορετικά συζητιόνται εκεί από ό,τι τα συζητάμε εδώ, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και υπάρχουν και τα γενικά ζητήματα. Από αυτά που είπαμε, και αξίζει να το ξαναπούμε, ότι πρέπει να δεχτούμε πως είναι ένα επιπλέον μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και γενικά όλοι το δεχόμαστε. Όμως πρέπει να τονίσουμε για αυτούς που είναι εδώ από την Κομισιόν για να το περάσουν το μήνυμα στην Κομισιόν, ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να αντιδρούμε σε καταστάσεις οι οποίες ε, προκύπτουν καθοδός στη ζωή μας. Εμείς θα θέλαμε να είχαμε καλύτερα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών και μυστικών πληροφοριών βασικά που να γίνονται γνωστές από τις μυστικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ασφάλειας πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνονται ήδη από την αρχή. Και από την άλλη μεριά δεν πρέπει να θεωρούνται ύποπτοι άνθρωποι οποίοι κάνουν κάποιες κρατήσεις στις μεταφορές. Περνάμε δύσκολους καιρού, αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα συμφέροντα των περισσότερων ανθρώπων. Πώς χειριζόμαστε τα προφίλ των επιβατών. Είναι πράγματα όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται πριν φτάσει ο καθένα στο αεροδρόμιο. Και άντε και φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Είχαμε τις ρυθμίσεις για τα υγρά, για τα παπούτσια, για τα πακέτα. Και αν καταφέραμε στην τελευταία αυτή περίπτωση και εντοπίσαμε τα παγιδευμένα πακέτα, ήταν επειδή ακριβώ είχαμε καλέ πληροφορίε. Από τι μυστικέ πληροφορίε ενημερωθήκαμε σωστά. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό. Οι υπηρεσίε ασφάλεια να κάνουν καλύτερα τη δουλειά του. Λοιπόν, όταν φτάσουμε στο αεροδρόμιο, πια Φτάνουμε στους αρρωτές σώματος. Στον Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε διαφορετική θέση από τους άλλους συναδέρφους. Τα επιβάλαμε εδώ και καιρό στο κοινό μας τα μηχανήματα αυτά. Ξέρω ότι και το Σκύπολ τα δοκίμασε και αυτά που είπε ο εισηγητής είναι πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχουν, υπάρχει αυτή η τεχνολογία με τα χιλιοστομετρικά κύματα. Υπάρχει επίσης και το software εκείνο που βασίζεται σε συστήματα επεξεργασίας εικόνας. Στο Χίθρο και στο Μάντσεστερ χρησιμοποιούμε την οπισθοδιάχυση των ακτίνων Χ. Η Επιτροπή θα ετοιμάσει κάτι και αυτό πρέπει να είναι κάτι που να μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, να υπάρξει κάποια αναρμόνιση. Πάντως συμφωνώ με τον εισηγητή για το ότι πρέπει να τονίσουμε την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας. Πολλές επιχειρήσεις και οργανώσεις έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας, ε, τα λόμπι, και υποστηρίζω απόλυτα εγώ αυτό που λέει ο εισηγητής, υπέρ των επιβατών δηλαδή. Τι μπορεί να κάνει ένα μηχάνημα δεν είναι μυστικό. Έχουμε το Wikipedia τελευταία. Ε, ξέρουμε τι γίνεται στα κομπιούτερ του Πενταγώνου. Όλοι περνάμε μέσα από τα μηχανήματα ανιχνευτών ε, μετάλλου. Μας ενδιαφέρει να μπορούμε να το πίσουμε ε, τα εκρηκτικά Υπάρχει τεχνολογία γι' αυτό. Άρα πρέπει να συνδυάσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πάντω σίγουρα στηρίζουμε αυτό το νέο μέσο, αλλά συγχρόνω πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να έχουμε στη διάθεσή μα την καλύτερη δυνατόν τεχνολογία. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονε για την υγεία που λένε ότι δεν είναι πρόβλημα για τους ανθρώπους που περνάνε από τα μηχανήματα πιστοδιάχυσης, περνάνε κάθε τόσο, αλλά πραγματικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο τους επιβάτες, αλλά και τους υπαλλήλου που δουλεύουν εκεί και οι οποίοι αναγκάζονται να περάσουν μέσα από σαρωτές σώματος, για παράδειγμα, πολλές φορές την ημέρα. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμπέρασμα. Όπω είπε και ο συγητή, θα υποβληθούν τροπολογίε και εγώ θα υποβάλω μια-δυο τροπολογίε για να τονίσω ακριβώς αυτά που σας είπα εδώ. Τελικά ελπίζω η Κομισιόν να μας ακούσει. Το ίδιο και τα κράτη-μέλη και έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κρι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω εκ μέρου ε, του κ. Ούτζια, που είναι ε, σκιώδη συγητή και σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών εκ μέρους του θέλω να πω ότι χαιρετίζει την έκθεση και θα περιμένει τις τροπολογίες. Συμφωνεί ότι οι σαρωτές σώματος δεν μπορεί να θεωρηθούν εντελώς αυλαβείς και πρέπει να το εξετάσουμε. Τώρα, ένα θέμα που πρέπει να συζητήσω και εγώ από ε, δικής μου προσωπικής ε, άποψη εκτός από του κοιόδους του. Όπω ε, ακούσαμε και από τη Jack Foster, ε, ακούσαμε ποιε είναι οι ε, διάφορε ανησυχίες και προδιαγραφές για τους αρρωτές σώματος. Υπάρχουν ανησυχίες ε, για ε, ε, επίπτωση επί του οργανισμού, όπως υπάρχουν και από τα κινητά τηλέφωνα. Αλλά αν φοβόμασταν οτιδήποτε δημιουργεί προβλήματα, ούτε θα οδηγούσαμε καν, γιατί ξέρουμε ότι από τα τροχαία ατυχήματα υπάρχουν πάρα πολλά θύματα κάθε χρόνο. Οτιδήποτε έχει τεχνολογία, αναγκαστικά μπορεί να έχει επιπτώσεις επί του πληθυσμού. Ε, φαντάζομαι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και οπουδήποτε αλλού, όταν εισάγεται μια νέα τεχνολογία, αν φανεί ότι είναι επιβλαβή, οι κατασκευαστέ και οι αρχέ των αεροδρομίων και οι κυβερνήσει θα διατρέχουν τον κίνδυνο να του καταγγείλουν και να ασκηθούν αγωγέ εναντίον του ε, για διάφορα θέματα. Και ο εξοπλισμό που θα απολύεται δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στου επιβάτε. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κοινό μέλημα και τα χρήματα που επενδύονται, επενδύονται προς μια κατεύθυνση που θα είναι αποδοτική. Δεν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Στην πρότασή μας εδώ αναφέρονται διάφορες τεχνολογίες. Δεν γνωρίζω τις διαφορές τεχνολογίες που αναφέρονται εδώ. Ούτε γνωρίζω τι συνέπειε από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι εμεί στο Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να επιλέξουμε τεχνολογίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσω πρέπει να θέσει όρια έκθεση και πιθανού κινδύνου και αν μπορεί η Επιτροπή να μας εξηγήσει πώς τίθενται αυτές οι προδιαγραφές θα ήμουν ε, ευτυχής. Είναι πρότυπα τα οποία τίθενται σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι προτάσεις υπάρχουν για του σαρωτέ σώματο, Ποια είναι η αρχή που χορηγεί άδειε για τέτοια θέματα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια αρχή που δίδει άδειε για εξοπλισμό που εκπέμπει ακτινοβολία. Από τις προτάσεις του εισηγητού δεν είναι σαφές για μένα Ποιο θα πρέπει να λάβει μέτρα και τι είδου μέτρα πρέπει να ληφθούν. Παραδείγματο χάρη στην παράγραφο 3 λέγεται, προτείνεται να αποφύγουμε αυτή την τεχνολογία. Να αποφύγουμε ποιοι είμαστε εμείς που θα αποφύγουμε για ολόκληρη την Ευρώπη, να απαγορευτεί δηλαδή αυτή η τεχνολογία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι ακριβώ ζητάμε με την έκθεση αυτή είναι, θα έπρεπε να είναι μια πρόταση που θα ζητάει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να διερευνήσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Δεν ξέρω λοιπόν αν η έκθεση αυτή αναφέρει κάποιες ανησυχίες για ορισμένες τεχνολογίες και όχι έναντι άλλων τεχνολογιών. Δεν πολύ καταλαβαίνω τι μας ζητάει να ψηφίσουμε. Είναι σαν να είμαστε σε ένα καφενείο και μεταξύ τυρού και αχλαδιού να λέμε «Α, δεν μας αρέσουν σε σώματος, να κάνουμε κάτι άλλο» θέλω να πω ότι δεν μου φαίνεται πολύ αντικειμενική αυτή η πρόταση που έχουμε ενωπιών μας. Um, Επίσης συνειδητοποιώ ότι τους τελευταίους μήνες περνάω από σαρωτές σώματος στο τοπικό μου αεροδρόμιο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μου κάνουν έλεγχο διαχειρός το προσωπικό ασφαλείας. Και φαντάζομαι ότι και εγώ χαίρομαι που δεν περνάω από αυτό το προσωπικό έλεγχο και το προσωπικό χαίρεται που δεν χρειάζεται να περνάει από έλεγχο κάθε επιβάτη. Άρα υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, εκτό από το βασικό που ανέφερε η Τζάκη Φώστα ότι αποφεύγουμε την τρομοκρατία, είναι και ότι πρακτικά ίσω είναι πιο ευχάριστοι οι σαρωτέ σώματος. Ευχαριστώ. Περιμένω τι απαντήσει τη Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Κρίς. Ευχαριστώ πολύ. Διαρωτώ με αν οι σαρωτέ σώματο όντω θα μα δώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί μπορούν να ελέγξουν μόνο την επιφάνεια του δέρματο, όχι αυτά τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σώμα ή σε πτυχέ του σώματο. Οι ακτίνε ε, ρόντγκεν, οι ακτίνε χι θα μπορούσαν να, τις, ε, να το ελέγξουν αυτό ε, υπάρχουν εκρηκτικά τα οποία μπορεί να κρύβονται σε πτυχές του σώματος και δεν ανοιχνεύονται από αυτούς τους ερωτές σώματος. Άρα τι χρησιμεύουν αυτοί οι ερωτές σώματος. Αν μπορεί κανείς να φέρει εκρηκτικά ε, τα οποία ε, δεν ανοιχνεύονται από τους ερωτές ε, που ανοιχνεύει μόνο την επιφάνεια του δέρματος, δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητα. Επίσης αναφέραμε το θέμα των επιπτώσεων επί της υγείας ε, επιβαρύνεται, ο οργανισμός από την ε, ακτινοβολία και στα χιλιοστομετρικά κύματα ε, είναι αντίστοιχη η ακτινοβολία όπως στα κινητά τηλέφωνα και στα μικροκύματα διάβασα και η Επιτροπή κάπου γράφει ότι είναι παρόμοια η ακτινοβολία όπως και στα κινητά τηλέφωνα και στα ε, κινητά τηλέφωνα πάλι γίνεται η συζήτηση για το κατά πόσο επιβαρύνεται ο πληθυσμό που τα χρησιμοποιεί. Υπάρχουν επίση τα θέματα που αφορούν τα παιδιά και τι εγγύου, αλλά και του ε, υπαλλήλου που συνεχώ εκτίθενται στην ακτινοβολία στα αεροδρόμια. Ε, είναι σημαντική και η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της, ε, του ιδιωτικού χώρου των ατόμων που ελέγχονται. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν μπορούν 100% να, να θεωρήσουμε ότι είναι εγγυημένη και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που μπορεί ε, να συμπεριλαμβάνουν προθέσεις ή καθετήρες ε, ή πάνες νομίζω ότι ε, δημιουργούν κινδύνους έκθεσης για αυτούς που ελέγχονται. Και θα πρέπει ε, ιδιαίτερα για τα παιδιά να φροντίσουμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τα αγγίζουν ξένοι και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ε, να εκτίθεται τα παιδιά σε κίνδυνο προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι και στα άλλα μέσα μεταφορών εξάλλου. Δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχουν ατυχήματα, τα χρησιμοποιούμε παρόλα αυτά νομίζω ότι στα αεροδρόμια που το χρησιμοποιούν ε, ε, έχουν γίνει πιο μεγάλες οι ουρές, δεν έχουν διευκολύνει ε, οι δοκιμές τουλάχιστον που γίνονται στις αεροτές σώματο, και εγώ θα προτιμούσα να το απορρίψουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Γιολάντα Χιούμπνερ. Mm, Ευχαριστώ πολύ. Υποτίθεται ότι με τους αρωτές αυτούς θα είχαμε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους επιβάτες των αεροπλάνων. Όμως θα πρέπει να σταθμίσουμε τα πράγματα. Πόσο μεγαλύτερη ασφάλεια θα έχουμε ε, με αυτούς τους αρωτές. Και από την άλλη πλευρά πόσο θα μας κοστίσουν αυτοί οι αρωτές όσον αφορά την υγεία των επιβατών. Διότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι τελείως υγιείς όλοι όσοι περνάνε αυτούς τους αρωτές. Κάποιος μπορεί να, είχε, να έκανε μια εγχείρηση, κάποιος άλλος μπορεί να έχει ένα βηματοδότη, μπορεί να έχει κάποια άλλα εξαρτήματα τέλος πάνω του πριν περάσει από τους αρωτές. Επομένως, οι σαρωτέ μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές παρενέργειες στην υγεία ενός ανθρώπου αν κάποιο έχει κάνει μια εγχείρηση, επαναλαμβάνω, δεν νομίζω θα του κάνουν καλό οι σαρωτέ. Κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων, δεν λέω. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα για τους επιβάτες. Δεν είναι μόνο τα παιδιά και οι έγκυες. Όλοι θα μπορούμε να επηρεαστούμε από την ακτινοβολία. Και προφανέ, προφανή θύματα. Προφανώ θα είναι τα, οι, οι, οι και τα παιδιά. Μία έγκυο, αν περάσει από αυτόν τον σαρωτή και δεχθεί αυτή την ακνοβολία, δεν ξέρουμε τι παρενέργειε θα έχει, τι συνέπειε θα έχει αυτή η ακνοβολία για το, για, στο έμβριο. Δεν ξέρουμε τι παιδί θα γεννήσει. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρουμε πόσο κακό μπορεί να κάνουν αυτέ οι ακνοβολίε στην ανθρώπινη υγεία. Όντω, ξέρουμε ότι οι τρομοκράτες μας, χρησιμο, μας ε, απειλούν και χρησιμοποιούν ούτε όχι μονάχα σε επίπεδο απειλή, αλλά και χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες, διάφορα τεχνάσματα τα οποία μας εκπλήσουν κάθε φορά. Και όντως συμφωνώ με την ε, συνάδελφο η οποία είπε προηγουμένως ότι θα πρέπει να στηριχθούμε σε μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών για τα πακέτα. Είδατε ότι όντως ε, λόγω της ε, της ε, καλής ενημέρωσης μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τον κίνδυνο. Άρα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε περισσότερο είναι καλύτερη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν είναι η πανάκια το να... οι σαρωτές, διότι είδαμε ότι οι σαρωτές κάνουν κακό στην υγεία. Δεν πρέπει να βιαστούμε επομένως. Δεν λέω ότι οι σαρωτές μπορεί να μην αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στο μέλλον, αλλά επί του παρόντος όμως δεν ξέρουμε ποιες είναι οι παρενέργειες των σαρωτών. Δεν ξέρουμε. Ευχαριστούμε, Κρήτον. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα και εγώ με τους συναδέλφους που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους. Πιστεύω επίσης, όπως είπε και η κυρία Γουίλσο πριν από λίγο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αν εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, την επόμενη φορά που ελπίζω να μην υπάρχει, κάποιος θα βρει έναν άλλο τρόπο να ξεπεράσει όλους αυτούς ε, τους ε, τρόπους που έχουμε εμείς εφεύρει για έλεγχο και να απειλήσει ανθρώπινες ε, ζωές. Πάντα θα συζητάμε δηλαδή για νέα τεχνολογία και ξανά νέα τεχνολογία και δεν θα τα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι να σταματήσουμε τις επιθέσεις. Δεν είναι αναλογικό αυτό το μέτρο και ανησυχώ πάρα πολύ για τις επιπτώσεις στην υγεία. Άκουσα τους κινδύνους και το γεγονός ότι σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούνται οι... τα μηχανήματα αυτά, δεν το καταλαβαίνω. Πώς είναι δυνατόν μερικές χώρες να χρησιμοποιούν αυτά τα μέτρα σε κάποια αεροδρόμια από που περνάνε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτοί που φεύγουν από τη χώρα, μπαίνουν στη χώρα. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα πριν καν μπούμε στη συζήτηση της επέκτασης των μέτρων αυτών. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή Υπάρχει τεχνολογία των ενεργών χιλιοστομετρικών κυμάτων και των παθητικών χιλιοστομετρικών κυμάτων που είναι και φθηνότερο σύστημα και δεν εκπέμπει ακτινοβολία καταγράφονται κάποια ε, σημεία του σώματος αλλά με μια θολή ε, ε, εικόνα και μπορούν να ανοιχνεύονται μεταλλικά και μεταλλικά αντικείμενα. Ενδεχομένως λοιπόν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την περισσότερη δηλαδή ακτινοβολία. Δεν είναι ασφαλής η μέθοδος που θα μπορούσε να ανοιχνεύσει αντικείμενα που βρίσκονται κρυμμένα σε πτυχές του σώματος. Εγώ απορρίπτω όλες τις, ε, όλα τα συστήματα ε, ενεργού ακτινοβολίας ε, είτε περιέχουν είτε αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν ακτίνες χ είτε άλλη ενεργό ακτινοβολία το μόνο που θα ήταν αποδεκτό θα ήταν τα παθητικά χιλιοστοματικά κύματα νομίζω ότι καταλήγουμε σε ένα διέξοδο γιατί ποτέ δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κάποιον να ε, προκαλέσει μια έκρηξη σε ένα αεροπλάνο. Νομίζω ότι είναι αδιέξοδο το να προσπαθούμε να αποφύγουμε κάθε πιθανό κίνδυνο θα μπορούσε κάποιος να έχει φάρμακα μαζί του και να κάνει ανάμιξη χημικών συστατικών, ανάμιξη πρώτων υλών ε, και να ανατινάξει το αεροσκάφος. Δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ασφάλεια. Νομίζω ότι ακόμη και στα tax free ε, μπορεί να βρει κανείς προϊόντα ε, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν προϊόντα σε ολόκληρο τον κόσμο που πολλούνται και μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς κατά τη διάρκεια της πτήσης. Θα έπρεπε τα tax free να τα έχουμε στο σημείο άφηξης του αεροσκάφους, ώστε να μην μπορεί κανείς να έχει μια φιάλη μαζί του για να αναμίξει τα διάφορα συστατικά. Ε, θέλω να πω ότι είναι αδιέξοδο το να προσπαθούμε να αποκλείσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Ούτε μπορούμε να βάλουμε τις ε, μυστικές υπηρεσίες ε, να ανοιχνεύουν με σερωτές σώματος κάθε πιθανό κίνδυνο. Αν δεν μπορούν οι τρομοκράτες να βρουν καμία λύση και τους έχουμε αποκλείσει κάθε κίνδυνο για αεροπειρατεία και ε, πρόκληση κινδύνου στους αεροσκάφη, θα επιλέξουν κάτι άλλο, σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σταθμούς του μετρό. Δεν θα μπορούμε πια να βγούμε από το σπίτι μας, αν νομίζουμε ότι μπορούμε να αποκλείσουμε τα πάντα. Είναι πραγματικά απαραίτητο να προσπαθούμε ε, να αποκλείσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο ε, τρομοκρατίας. Καλύτερη, νομίζω, προσέγγιση θα ήταν μια ανοιχτή κοινωνία. Εγώ απορρίπτω όλα αυτά τα μέτρα, είναι δαπανηρά, ε, προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και, ε, και τα προσωπικά δεδομένα και δεν αποτελούν και λύση. μπορούμε να δούμε από τις αναλύσεις της Επιτροπής και καλό θα ήταν να κάνει η Επιτροπή της αναλύσεις του τι είναι αποτελεσματικό από αυτά τα μέτρα κατά πολέμηση της τρομοκρατίας. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα αφήνουμε να περνάνε τέτοιες μέθοδοι που προσβάλλουν την προσωπική αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας ήμουν στις μεταφορές που ψηφίζαμε, γι' αυτό άργησα. Θέλω να σας πω ότι για τις αρωτές σώματος η βασική πτυχή το λένε και το συζητάμε και με τους ειδικού, είναι η αύξηση της ασφάλειας σε έναν τομέα όπου η ασφάλεια είναι πολύ βασική για να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί ελεύθερα, όπως είναι οι επιβάτες ενέργειες μεταφορές. Μιλήσαμε λοιπόν για τη δυνατότητα αυτή χρήσης των σαρωτών σώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια, για προστασία συγχρόνως της υγείας, αλλά και για ε, να αισθάνεται πιο άνετο επιβάτη, ο οποίο δεν αισθάνεται πάντα καλά όταν έρχονται οι υπάλληλοι και ψηλαφίζουν το σώμα του για να τον ελέγξουν. Αν υπάρχουν μηχανισμοί λοιπόν, αν υπάρχει τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτούς τους στόχους, τότε πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε όπως κάνουμε και με άλλες τεχνολογίες για αντίστοιχους λόγους. Αλλά πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, εννοείται. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας πρέπει να τις θέσει αυτές τις προϋποθέσεις. Υγεία πρώτα απ' όλα. Από τις διάφορες παρουσιάσεις που είχαμε από ειδικού, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούν να μας εγγυθούν 100% ότι μια τεχνολογία είναι αυλαβής, για παράδειγμα, για τους εργαζόμενους, είτε είναι οι πιλότοι, είτε είναι το προσωπικό στα αεροπλάνα, στα αεροδρόμια που περνάνε συχνά από τα μηχανήματα αυτά ή οι επιβάτες που ταξιδεύουν πολύ συχνά και άρα περνάνε πολύ συχνά από τους ερωτές αυτούς. Σίγουρα στη ζωή μας πολλές φορές ε, έχουμε ακτινοβολία με διάφορους τρόπους. Ε, αν μη τι άλλο, εδώ πέρα να ζητήσουμε εγγύσεις για την ασφάλεια, ώστε αυτοί που ταξιδεύουν πιο συχνά ή το προσωπικό που δουλεύει επιτόπου στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα να μην κινδυνεύει. Εμένα αυτό που με ενοχλεί όταν πήγα για παράδειγμα σε ένα αεροδρόμιο που τους είχε τους ερωτές αυτούς, δεν με ρώτησαν, στο Βούργο, δεν με ρώτησαν θέλετε ή δεν θέλετε, μου τα επέβαλαν. το θέμα της ανάλυσης εικόνων. Το είδαμε και στις Ηνωμένε Πολιτείε πρόσφατα ότι δεν ξέρουμε 100% αν είναι σίγουρα τα μηχανήματα αυτά. Έπειτα, το θέμα του κόστους και της αποτελεσματικότητας. Αυτή η σχέση πρέπει να μελετηθεί, γιατί κοστίζει ακριβά η τεχνολογία αυτή αν το Κοινοβούλιο συζητάει υποχρεωτική ή μη υποχρεωτική αυτή η τεχνολογία, πριν καταλήξουμε να λάβουμε υπόψη μας το κόστος. Πάντως, επαναλαμβάνω, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την ασφάλεια των μηχανημάτων αυτών. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή γιατί έχει ιεραρχήσει πολύ καλά τις προτεραιότητες στο κείμενό του. Εν συντομία, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις ανησυχίες για την υγεία, να πω ότι περνάω σαρωτές κάθε εβδομάδα δεν, και δεν έχω πεθάνει ακόμα, δεν είναι άμεσος ο θάνατος. Μήπως θα μπορούσε η Κομισιόν να μας απαντήσει στα θέματα υγείας, δηλαδή ε, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής ε, για την... Ε, για τις παρενέργειες στην υγεία των επιβατών. Ο κύριος Περιό, κοιτάξτε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Ριβελίνη για την ε, έκθεση που μας έκανε και για τις προτάσεις αυτές. Θέτει μια σειρά ερωτήσεων ε, που πρέπει όντως ε, να τις εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς ζητάμε όλο ένα και περισσότερο ασφαλή αεροδρόμια. Αεροδρόμια ε, όπου θέλουμε ο έλεγχος να είναι πιο γρήγορος, ε, πιο εύκολος ενδεχόμενα. Ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγξαν και στη Βουδαπέστη και στην Ιταλία. Από ό,τι φαίνεται τα συστήματα ελέγχου δεν ήταν ε, αρκετά ασφαλή. Επίσης για τα θέματα της υγείας. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε λειτουργία ένα ε, εργαλείο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Επομένως, είναι απαραίτητο το εργαλείο αυτό να είναι ασφαλές. Η έλεγχη πρέπει να είναι ασφαλής προφανή, προφανώς, αλλά θα πρέπει να μην ε, βλάπτουν την υγεία. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ακούστηκαν πολλές απόψεις, αλλά όλοι θέλουμε οι, οι έλεγχοι να γίνονται πιο γρήγορα, όλοι είμαστε επιβάτες. Ε, ε, αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, γι' αυτό θα ήθελα ο Ριβελίνη να το λάβει και αυτό υπόψη του. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φώστερ που την, ε, τον ξαναζήτησε. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο να κάνω στον συνάδελφο Chris Ντέιβις. Ε, κανείς δεν ε, διασκεδάζει με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε μια προοπτική. Εγώ 20 χρόνια δούλεψα στα, στις, ε, αεροπλάνα, έχω δει τα πάντα, έχω διαβάσει βιβλία, έχω δει ταινίε και τα λοιπά για την ασφάλεια. Επομένω, το τελευταίο άτομο που θα λάβει, θα όλα αυτά τα πράγματα έτσι ελαφρά την καρδία. Όμως θέλουμε να έχουμε ένα συμπληρωματικό εργαλείο, αν θέλετε, για να ε, καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Το δεχόμαστε και η γνώμη το δέχεται. Αλλά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία, το ξέρουμε ότι είναι διαθέσιμη αυτή η τεχνολογία, που είναι λιγότερο βλαβερή από κάποια άλλη τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιείται. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτό συζητάμε. Επίσης, δεν λέμε, ε, λέμε ότι δεν μπορεί η Κομισιόν να μας λέει, να μας επιβάλλει τι τεχνολογία θα χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να δημιουργηθεί απλώς ένα πλαίσιο έτσι ώστε να υπάρχει μια κάποια ε, ε, ε ομοιομορφία στην Ευρώπη. Δεν περνάς αυτή τη στιγμή συνέχεια σαρωτές, ε, τυχαία σε επιλέγουν για να περάσεις. Όμως αυτό το οποίο λέμε, επί παρόντος τουλάχιστον, λέμε όμως ότι υπάρχουν και μέλη του προσωπικού τα οποία περνάνε συνέχεια και κάποιοι ε, ε, συχνοί επιβάτες και δεν ξέρουμε ακόμα τις παρενέργειες διότι δύο μήνες χρησιμοποιούνται. Επομένως, ε, θα πρέπει να δούμε και μακροπρόθεσμα τι γίνεται. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν, αλλά θα πρέπει να είμαστε ε, ρεαλιστές. Να χρησιμοποιήσουμε την βέλτιστη δυνατή τεχνολογία και να χρησιμοποιήσουμε και τα ε, άλλα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα, μυστικέ υπηρεσίε, ανταλλαγή προφοριών κτλ. για να προστατευτούμε. Και α είμαστε ενήλικοι, σα μιλάμε σοβαρά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ να δώσω το λόγο στον κύριο Φιλίπ Κονέλης για την Επιτροπή. Τρία-τέσσερα λεπτά όμως, αν είναι εύκολο, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ριβελίνη για το σχέδιο γνωμοδότησης που είναι πολύ συγκεκριμένο και θέτει επιτάπητος ε, τα πραγματικά ζητήματα που θα μας βοηθήσουν πολύ στο έργο μας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση λοιπόν σήμερα το πρωί. Επίσης θέλω να σας ε, πω ότι ε, ε, δουλεύουμε για την αξιολόγηση επιπτώσεων. Αρχίσαμε την αξιολόγηση επιπτώσεων πριν από λίγους μήνες και ελπίζουμε ότι θα το ολοκληρώσουμε μέσα στις προσεχείς εβδομάδες. Σήμερα λοιπόν είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση γιατί έχουμε μια αρχική εντύπωση για την θέση της Επιτροπής σας. Στην αξιολόγηση επιπτώσεων εξετάζουμε τα συνήθεια, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κλπ. Και αυτή η αξιολόγηση επιπτώσεων, κοινωνική επίπτωση παραδείγματο χάρη, είναι πολύ σημαντική δεδομένων των ε, επιπτώσεων επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των επιπτώσεων επί της υγείας. Και θα αφιερώσουμε μεγάλο μέρος της αξιολόγησης επιπτώσεων στις επιπτώσεις επί, την, επί μια γενική παρατήρηση τώρα θα ήθελα να αναφέρω ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν τέλεια μηχανήματα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για την ασφάλεια της αεροπλοείας. Όλες οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες έχουν μειονεκτήματα μερικές φορές μειονεκτήματα ασφαλείας, μερικές φορές ε, πρακτικά μειονεκτήματα, πρακτικές δυσκολίες για τους επιβάτες. Αλλά όταν έχουμε μια απειλή για την πολιτική αεροπορία και όταν θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μέτρα προστασίας, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για να γίνεται κάποιο έλεγχος των επιβατών και του προσωπικού. Η καλύτερη εφικτή λύση που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι ανάγκε που έχουμε, δηλαδή επαρκέ επίπεδο ασφαλείας και ω το δυνατόν καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Για θέματα υγείας τώρα πιο συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση επιπτώσεων, όπως είπε ο εισηγητής, θα κάνουμε διάκριση μεταξύ της τεχνολογίας χιλιομετρικών κυμάτων και της τεχνολογίας ιονίζωσης ακτινοβολίας. Και αυτό που μπορώ να πω προς το παρόν ε, γενικά για τα χιλιοστομετρικά κύματα και στις δύο περιπτώσεις ε, μπορούμε να βασιστούμε σε υφιστάμενους κανόνες ε, και εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα χιλιοστομετρικά κύματα τα γενικά μας ευρήματα είναι όπως και σε άλλες εφαρμογές όπως κινητά τηλέφωνα ή φούρνους μικροκυμάτων. Το κύριο ζήτημα είναι η ένταση της έκθεσης στην ακτινοβολία γιατί δεν υπάρχει σωρευτική έκθεση αντίθετα με αυτό που ισχύει για την ιονίζουσα ακτινοβολία. Θα ήθελα να πω λοιπόν ως γενικό σχόλιο ότι εφόσον η ένταση της ακτινοβολίας δεν είναι υψηλή όταν περνάμε από ένα σαρωτή, κανονικά δεν υπάρχουν προβλήματα για την υγεία. Αυτό μας έχουν πει οι εμπειρογνώμονες. Για την ιονίζουσα ακτινοβολία, πάλι μπορούμε να βασιζόμαστε στην υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία από ακτινοβολία σύμφωνα με τη συνθήκη Ευρατόμ που αφορά κάθε είδος έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία για μη ιατρικούς σκοπούς και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιου είδους ακτινοβολία και οι σωματεία σώματος δεν θα είναι η τελευταία περίπτωση στην οποία εφαρμόζουμε τέτοια νομοθεσία. Οι γενικές αρχές αυτής της υφιστάμενης νομοθεσίας έχουν τρία σκέλη. Καταρχήν, η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας για μη ιατρικούς σκοπούς θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και οτιδήποτε ενέχει έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία πρέπει να είναι αιτιολογημένο, ούτω ώστε να είναι σαφής, σαφές το όφελος προς το άτομο και προς την κοινωνία, ε, χωρίς να υπάρχουν ε, ε, υψηλότερες δυσμενείς επιπτώσεις από τις θετικές επιπτώσεις. Ε, δεύτερον, θα πρέπει η προστασία της υγείας να είναι βελτιστοποιημένη, ώστε οι δόσεις να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Και τρίτον, οι δόσεις ακτινοβολίας πρέπει να είναι περιορισμένες για να διασφαλίσουμε ότι κανένα άτομο δεν θα εκτίθεται σε δόση πάνω από την ε, νομικά ισχύουσα δόση ακτινοβολίας. Και πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν μια αρχή προστασία από την ε, ιονίζουσα Ακτινοβολία που θα εξετάζει τα θέματα αυτά και θα καταλήγει σε γνωμοδότηση για το εφικτό και για τι προποθέσει που θα ισχύουν για τον εξοπλισμό που εκπέμπει η ιονίζουσα Ακτινοβολία. Στο παρόν στάδιο λοιπόν αυτά μπορώ να σας πω για τα δικά μας ευρήματα κατά την αξιολόγηση επιπτώσεων που όπως σας είπα μέσα στις προσεχείς εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε μπορούμε και να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, αν θέλετε, και να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ένα λεπτό, ε. όχι παραπάνω. Ευχαριστώ. Ήμασταν στο ΣΥΠΟΛ τις προάλλες και εκεί χρησιμοποιούν τους σαρωτές, έχουν πέντε χρόνια εμπειρία. Πολλοί υπάλληλοι περνάνε πολλές φορές την ημέρα από τα μηχανήματα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί παρακολουθούνται ιατρικά. Ακριβώς γιατί αυτοί είναι που χρησιμοποιούν περισσότερο τα μηχανήματα. Μετά από πέντε χρόνια λοιπόν δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα υγείας στους ανθρώπους αυτούς που περνούν, όπως σας είπα, πολλές φορές καθημερινά από τα μηχανήματα αυτά. Πέντε χρόνια. Πήγα κι εγώ στο Σιμπολβόλ και πέρασα κι εγώ από τα μηχανήματα αυτά. Απλώς αυτό δεν θέλω να σας πω, να σας ενημερώσω. Καλώς. Κοιτάξτε, ωραία, μπορείτε και γραπτά να μου απαντήσετε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γιατί πόσο κοστίζουν τα μέτρα αυτά και γιατί δεν συζητάμε λίγο και για τη μεταφορά της απειλής σε άλλες μορφές ε, μεταφορών. Γιατί δεν το κάνετε αυτό καθόλου. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε όλα αυτά, αλλά γραπτά. Δεν πειράζει, γραπτά. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εκτός μικροφώνου η Πρόεδρος. Πρόκειται για μία έκθεση που από ό,τι είδαμε ενδιαφέρει πάρα πολύ τους συναδέρφους. Οπότε κύριε Σιγητά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Πραγματικά στράφηκε πολύ η προσοχή ε, μας σε αυτή την έκθεση. Εμείς είμαστε αιρετοί νομοθέτες, αν θέλετε. Είμαστε υποχρεωμένοι να νομοθετήσουμε έτσι ώστε να υπάρχουν ισορροπημένες διατάξεις που να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Ποια δικαιώματα. Δικαιώματα υγείας εδώ. Δεν είναι μονάχα οι ακτίνες χ αν θα περάσουν τους ορωτέ, αλλά είναι και το δικαίωμα του επιβάτη, του πολίτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ταξιδέψει και ο οποίος ψυχολογικά θεωρεί ότι προστατεύεται από αυτά τα νέα τεχνολογικά μέσα θα πρέπει να διαφυλάξουμε και την ψυχολογική υγεία του ε, πολίτη. Το δικαίωμα μετακίνησης, το δικαίωμα ασφάλειας. Εμείς που είμαστε οι νομοθέτες, οι αιρετοί νομοθέτες, έχουμε το, την, ε, την, ε, την υποχρέωση να εξετάσουμε ισορροπημένα όλες αυτές τις προτάσεις και να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε διατάξεις οι οποίες να είναι ισορροπημένες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και απαντώ και στον συνάδελφο ο οποίος με ρώτησε τι κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Ε, τι θα ψηφίσουμε τέλος πάντων. Εγώ προσπάθησα να παρουσιάσω, με μεγάλη μετριοφροσύνη βέβαια, μία σειρά προτάσεων όπου ένα συγκεκριμένο σημείο προτα... προτείνω στους συναδέλφους να απαγορεύσουμε, να αποκλείσουμε τις ακτίνες Χ. Αυτό είναι σαφές στην έκθεσή μου, ότι η τεχνολογία αυτή των ακτίνων Χ δεν είναι η κατάλληλη και βλάπτει την υγεία. Και εδώ επανέρχομαι σε αυτά που λέει η Κομισιόν, στην έκθεση της Κομισιόν. Θα πρέπει να ισορροπήσουμε όλα τα δικαιώματα, θα πρέπει να προσφέρουμε την, ε, ε, την καλύτερη, την βέλτιστη ε, τεχνολογία που υπάρχει και βέβαια να την προσαρμόσουμε ανάλογα στο μέλλον, εάν και εφόσον υπάρχει κάποια άλλη πρόοδος. Και να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου Υπενθυμίζοντα όλα όσα είπε, έλεγε ένα φιλόσοφος για τις παραδόσεις, γιατί ήταν υπέρ των παραδόσεων, είπε ότι η... ο... ο σύγχρονος κόσμος, το, μοντέρνο, είναι ένα σπαθί. Εάν το πιάσεις από τη λαβή, πολύ καλά θα κάνεις. Θα, θα, μπορέσεις να υπερασπίσεις τον, τον εαυτό σου. Αν το πάρεις όμως από την άλλη πλευρά, από την ανάποδη, θα κάνεις κακό στον εαυτό σου. Το ίδιο είναι και η τεχνολογία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 6 Δεκεμβρίου του 2010, 12 ε, η ώρα. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα τον Απρίλιο και θα περάσει από την Ολομέλεια τον Μάιο. Περνάμε τώρα στο δεύτερο σημείο της ημερησίας διάταξης και αυτό πάρα πολύ σημαντικό σημείο που αφορά το, την έλλειψη πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η λύση σε ένα μακροπρόβλημα το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω τον λόγο... Συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον εισηγητή καταρχάς, Ξάμπα Σάντορ Ταμπατζή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια μεγάλη έλλειψη που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει να αυξήσει την παραγωγή ζωοτροφές με πρωτεΐνες ή να εισάγει κρέας από το εξωτερικό. Γι' αυτό το δίλημα Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολλές πτυχέ που έχουν να κάνουν τόσο με την υγεία όσο και με το περιβάλλον. Σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται όλο και περισσότερο στο έλεος των εισαγωγών. Οι ζωοτροφές, οι πρωτεϊνούχες, εισάγονται σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες. Συγχρόνως οι ανάγκες της Κίνας έχουν αυξηθεί Πράγμα που σημαίνει ότι στην παγκόσμια αγορά η Κίνα είναι μεγάλος ανταγωνιστής μας όσον αφορά την αγορά πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. Ε, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις πρωτεΐνες που έρχονται από ζωικές πηγές και τις πρωτεΐνες που έχουμε από φυτικές πηγές. Όσον αφορά της ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες. Η Dagmarot Μπέρεντ είναι η ειδική γι' αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μετά από την σπογκώδη κεφαλοπάθεια των βοηδών, το 96 δηλαδή, για τα μυρικαστικά, απαγορεύτηκαν πλήρως οι ζωοτροφές αυτές που περιέχουν ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες. Είναι ένα θέμα που έγινε ταμπού και εξακολουθεί να είναι ταμπού. Συγχρόνως όμως, οι ζωικές πρωτεΐνες έχουν ε, διαφορετικές ε, επιπτώσεις πάνω σε ζώα που δεν είναι μυρικαστικά. Η έκθεση Χάισλιν δεν το συμπεριλαμβάνει αυτό όμως. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν με τα μη μυρικαστικά? Ποια πρέπει να είναι η θέση μας για τις δικές τους ζωοτροφές στο μέλλον? Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη και να δούμε στην περίπτωση των ζώων που δεν είναι μυρικαστικά υπάρχει δυνατότητα να τους δίνουμε ε, ζωικές ε, πρωτεΐνες ή υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία. Θα δείτε ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι πολύ περιορισμένες όσον αφορά τις ε, ζωοτροφές που περιλαμβάνουν φυτικές πρωτεΐνες. Για λόγους τόσο κλιματικούς όσο και οικονομικούς. Όσον αφορά τους οικονομικούς λόγους, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ε, παραγωγή δημητριακών όσον αφορά την τιμή τους για παράδειγμα. Στη χώρα μου, την Ουγγαρία για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να καλλιεργήσει σόγια ή άλλα φυτά που χρησιμοποιούνται στις ζώτροφες δεν έχει κέρδος. Ενώ αν βάλει δημητριακά θα έχει 600 ευρώ κέρδος ανά εκτάριο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση γιατί δεν εχει κερδος ενω αν βαλει δημητριακα θα εχει 600 ευρω κερδος ανεκτάριο. καταλαβαινετε ποσο δυσκολη ειναι η κατασταση γιατι δεν μπορω να φανταστώ κάποιον που να μπορεί να κερδίσει παραπάνω 600 ευρώ και να μην θέλει. Γι' αυτό λοιπόν και οι γεωργοί το αποφεύγουν. Στη Γαλλία έχουμε παραδείγματα με την κοινή γεωργική πολιτική εξαιτία της αποσύνδεσης είναι πολύ δύσκολο να έχουν οι γεωργοί ενισχύσεις. Και έπειτα υπάρχει και άλλη πτυχή όπως σας είπα, η πτυχή περιβάλλον. η παραγωγή των ε, φυτικών ε, πρωτεϊνούχων ε, καλλιεργιών, σόγια, αραβόσιτος, δεν έχουν πρωτεΐνη μεν, αλλά τα παράγωγά τους έχουν υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεΐνης. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία να μπορέσουμε να ευνοήσουμε την παραγωγή ορισμένων προϊόντων που έχουν ως βάση την πρωτεΐνη και έτσι να μειώσουμε και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να περιορίσουμε την χρήση των λιπασμάτων, που αλλιώς είναι αναγκαία. Άρα λοιπόν για το περιβάλλον οι φυτικές αυτές ε, πρωτενούχες καλλιέργειες είναι πολύ σημαντικές χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες μας σε ζωοτροφές έτσι. Όταν εισάγουμε τέτοιες ζωοτροφές, πρέπει να ξέρουμε ότι πρόκειται για γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Άρα και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το ένα δέκατο των αναγκών μας το εισάγουμε ενώ η συγκέντρωση σε πρωτοΐνη είναι 25% σε εμά και τα 3 τέταρτα τα εισάγουμε. Και τα 2 τρίτα από τις εισαγωγές μας αυτές είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Και για να σας σοκάρω λίγο, πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μείγματα που κυκλοφορούν περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε ένα ποσοστό πάνω από 90%. Άρα, οι ελλείψεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη όσον αφορά τις ε, πρωτεΐνες δημιουργούν τεράστια προβλήματα τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία μας. Εξού και η πρότασή μου. Προτείνω στην μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής να στηρίξουμε την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνούχων προϊόντων, να ελέγξουμε πολύ περισσότερο τι γίνεται με τις εισαγόμενες ζωοτροφές, τις πρωτεϊνούχες, γιατί υπάρχει εδώ τεράστιος κίνδυνος. Προς το παρόν δεν έχουμε λύση και είμαστε υποκριτές, γιατί πολλοί λένε ότι είναι κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη τους ότι 90% τη εισακόμενη εισόγεια είναι γενετικά τροποποιημένη, ότι άρα οι ζωοτροφές που δίνουμε στα ζώα μας είναι με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κατά 90% και παραπάνω. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τέλος. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και να ζητήσω εδώ και την στήριξη ολόκληρης της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, για το εξή. Μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα αν αρχίσουμε να παράγουμε εμείς ε, φυτικές πρωτενούχες καλλιέργειες. Έτσι διευκολύνεται και η βιοπικιλότητα. Στην μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να το προσέξουμε αυτό πολύ. Επί του παρόντος δεν γνωρίζουμε τις τιμές Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να επιτρέψουμε την βιοπικιλότητα η οποία θα βοηθήσει να καταπολεμήσουμε και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό είναι αναγνωρισμένο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και αυτά προσπάθησα και να συμπεριλάβω στη γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Τώρα, μια που είμαι σκιώδης, θα πω δύο λόγια και εγώ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την ποιότητα της έκθεσής σας που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα που μπορεί για πολλούς να φαίνεται τεχνικό, αλλά άπτεται πολλών και διαφορετικών τομέων. Αναφερθήκατε στην ε, αυτάρκειά μας όσον αφορά τα τρόφιμα. Αναφερθήκατε στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εγώ θα προσθέσω εδώ ότι έχει να κάνει και με το δικό μας διατροφικό μοντέλο. Γιατί υπερκαταναλώνουμε κρέας. Και το γεγονός ότι η υπερκατανάλωση αυτή έχει να κάνει και με την παχυσαρκία, υπενθυμίζω ότι 6 με 36%. 160 εκατομμύρια ε, υπέρβαροι υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεν λέω ότι φταίει το κρέας, αλλά ότι πρόκειται για ένα διατροφικό μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει και το οποίο επηρεάζει η σόγια ε, για την οποία μιλάμε απευθύνεται για κατανάλωση από τα ζώα, όχι από τους ανθρώπους. Από το 1990 μέχρι το 2007 αυξήθηκε η κατανάλωση κρέατος κατά 5% στον κόσμο. Αυτό δημιουργεί και περιβαλλοντικά προβλήματα που τα συζητάμε συχνά. Υπάρχει η αποψήλωση των δασών η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνη για το μισό των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου και εκπέμπει περισσότερα τέτοια αέρια από ότι οι μεταφορές. Άρα εμείς που είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντος, που καθημερινά ασχολούμαστε με το κλίμα, πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Η αποψήλωση των δάσων επίση 20% των αερίων. Στην Αργεντινή τα τελευταία χρόνια πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια ε, δάσων καταστράφηκαν για σόγια. Και αλλού 86% της επιφάνειας του Ηνωμένου Βασιλείου περίπου 54% στην Αργεντινή των αρρώσιμων γιών. Τέσσερις φορές ε, οι κάτω χώρες και στον Αμαζόνιο. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό δασών θα καταστραφεί για να καλλιεργηθεί εκεί η σόγια. Δεν μπορεί λοιπόν το θέμα αυτό των πρωτεϊνών να το συζητάμε χωρίς να το βάζουμε σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τον εισηγητή μας, ο οποίος μας τα υπενθύμησε όλα αυτά. Υπάρχουν δύο πραγματάκια που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Το ένα είναι το ΜΕΓΑ Αυτό είναι ένα ζήτημα που μπαίνει όλο και περισσότερο. Γιατί το κρέας ζώων που τρέφονται με σόγια έχουν χαμηλά ποσοστά ποσοστά 3. Και αυτό μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα υγείας. Είναι ένα καινούριο θέμα που έχει τεθεί επιτάπητος. Σήμερα το πρωί όλο για υγεία μιλάμε. Το θέμα του γλυφοσάτ επίσης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία μας. Αυτά είχα να προσθέσω. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην Τάκμα Ροτ Πέρεν. Α, ποιος άλλος ζήτησε το λόγο? Η Τάκμαρ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ακούω τη συζήτηση και είναι σαν να την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση για πολλά θέματα και πολλές φορές. Καταρχήν, έντονες συζητήσεις έχουμε κάνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και 13 χρόνια. Πριν από 15 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούσαμε το θέμα της πογκόδους εγκεφαλοπάθειας των βοηδών. Από το 1997 έχουμε μια επιτροπή εξέτασης και μια ε, επιτροπή ε, παρακολούθησης δύο χρόνια αργότερα και είμαι και εγώ πρόεδρος της επιτροπής και με άλλους συναδέλφους ε, μεταξύ αυτών πολλοί δεν είναι πλέον ευρωβουλευτέ, ασχοληθήκαμε με το θέμα και νομίζω ότι το έχουμε παρακολουθήσει επαρκώ το θέμα. Τα γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα αυτά. Συζητάμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο εμείς δημιουργήσαμε και πρέπει ξεκάθαρα να δούμε ότι εμείς δημιουργήσαμε το πρόβλημα. Ο κ. Σταμπάτσης στην ε, παρέμβασή του μίλησε για την Επιτροπή Γεωργίας ε, ε, που σίγουρα θα δώσει μια καλή έκθεση. Πρέπει να πω ότι η έκθεση του εισηγητού του κυρίου Χόισλινγκ στην Επιτροπή Γεωργίας είναι εξαιρετική δύσκολα θα μπορούσε να γίνει καλύτερη αυτή η έκθεση. Εμείς βέβαια θα τη βελτιώσουμε, θα το προσπαθήσουμε. Ο κ. Σταπάτζης στην ε, παρέμβαση του πολύ καλά μας παρουσίασε την εξέλιξη σε σχέση με τον τομέα των πρωτεϊνών στη διατροφή των ζώων. Το θέμα που μας απασχολεί δηλαδή σήμερα. Και ένας συνάδελφός μου ε, που είναι αγρότης και είναι εκπρόσωπος των Πρασίνων Δυστυχώς δεν είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Φρίντριχ Γκρέφετ Σουμπάρινγκτορφ. Το είχε επισημάνει αυτό το θέμα πολύ νωρίς, ότι ε, με τα συναισθήματα δύσκολα κάνουμε καλή πολιτική. Γιατί μιλάμε για τις ζωοτροφές και για τη διατροφή των ζώων που έγινε πολύ ευαίσθητο θέμα και δημιουργεί συναισθηματική φόρτιση. Και ενθουσιαστήκαμε στο Κοινοβούλιο προς διάφορες κατευθύνσεις. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα και ο συνάδελφος ο Γκρέφε Τσουμπάριγκορφ ποτέ δεν το είχε καταλάβει και διαβάζοντας και την έκθεση Χόισλινγκ σήμερα νομίζω ότι στο σημείο 7 της έκθεσής του και αυτός ε, ε, όπως και ο κ. Τζαμπατζής στο σημείο 6 της γνωμοδότησής του ε, θέτει αυτό το θέμα της πηγής ζωικών πρωτεϊνών που πρέπει να το επανεξετάσουμε. Ναι, βεβαίως, συμφωνώ ότι πρέπει ε, να έχουμε πηγές πρωτεϊνών και να καλλιεργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τέτοια φυτά. Αυτό θα μας ανεξαρτητοποιήσει από τις εισαγωγές και θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε και την ποιότητα. Και δεν εννοώ μόνο για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, γιατί αυτό δεν το θέλουμε. Ξάλλου εγώ πάντοτε το έλεγα. Έλεγα να απαγορεύσετε ε, την κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών και την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένη σόγια στα ζώα. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Εδώ μιλάμε για φυτικά που είναι πρωτεϊνούχες καλλιέργειε και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξουμε. Όμω πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ποτέ δεν θα κατορθώσουμε για το ζωικό κεφάλαιο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε αυτάρκεις ε, σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Εκτός αν θέλουμε να έχουμε μόνο καλλιέργεια. Για την αναλλαγή των καλλιεργειών, πολύ σωστά τα λέει ο κύριο Χόισλινγκ και νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει. Λέμε ότι δεν θέλουμε εισαγωγέ ή θέλουμε λιγότερε εισαγωγέ. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε λοιπόν το θέμα των ζωοτροφών. Στο σημείο 6 του κυρίου Ταμπάτζη και στο σημείο 7 του κυρίου Χόισλινγκ βλέπουμε θέματα που πρέπει να απασχολήσουν την Επιτροπή. Η Επιτροπή τα ασχολείται με τα θέματα αυτά μόνο όταν φτάσει σε πρόβλημα, μόνο όταν ε, έχει οξυνθεί το πρόβλημα. Πρέπει να δούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ε, αν ε, εξετάσουμε το θέμα της διατροφής των μυρικαστικών, πάντοτε ήταν απαγορευμένο να τους χορηγούμε ζωικές πρωτεΐνες. οι κτηνοτρόφοι δεν το γνώριζαν ότι είχαν αναμειχθεί ζωικές πρωτεΐνες στις ε, φυτικές ζωοτροφές που έδιναν στα μυρικαστικά ή αν το γνώριζαν ε, τουλάχιστον δεν το παραδέχονταν. Επίσης δεν είναι δεοντολογικό ούτε αλεύρα να δίνουμε στα μυρικαστικά. Το περιορίσαμε στα ε, βοηδή ε, και στα νέα μοσχάρια, αλλά ε, όλοι ε, που βρίσκονται στα παράλια της Βαλτικής και στις ε, σκανδιναβικές χώρες ε, δεν μπορούν να θεωρούν εναλλακτική λύση το να ταΐζουμε με ηχθιάλευρα γεμάτα διοξίνες τα μυρικαστικά. Θα μου πείτε ποια είναι η εναλλακτική λύση. Αν αφήσουμε απ' έξω τα μυρικαστικά, γιατί δεν τίθεται θέμα για τα μυρικαστικά, μας μένουν αυτά τα ζώα που τρώνε τα πάντα, δηλαδή τα οι ε, και τα πουλερικά, που ε, ε, τρώνε τα πάντα, που είναι πανφάγα. Κατά τη σφαγή των ζώων θα πρέπει να δούμε αν έχουμε την πολυτέλεια να επιλέγουμε μόνο τα καλύτερα ζώα και να δούμε ποια είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και ποια είναι αυτά τα οποία δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, οπότε θα πρέπει να καταστρέφονται. Ξέρω ότι πρέπει να έχουμε την, πολιτέλη, την πολυτέλεια για να πούμε ότι δεν θα δώσουμε οποιαδήποτε ζωοτροφή ε, στα πανφάγα ζώα. Και ακούσαμε τι είπαν και άλλοι συνάδελφοι, είπαμε ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε κανιβαλισμό για τις ζωοτροφές. Και το καταλαβαίνω, τα ζωικά απόβλητα δεν μπορούμε να τα ταΐζουμε στα ζώα του ιδίου είδους. Τι να κάνουμε στο στο ίδιο ζώο πρέπει να δούμε ε, ε, ε, τι, ε, τι καταναλώνεται. Καταναλώνουμε το φιλέτο και το διπλανό κρέας είναι για πέταμα, οπότε τι θα το κάνουμε, το κάνουμε κρεατάλευρο. Πρέπει να εξετάσουμε και μικροβιολογικά τα προϊόντα με τον Γκρέφτσου Μπάλιντορφ και τον κύριο είχαμε ζητήσει να διαμορφωθεί μια μέθοδος που συμπεριλαμβάνει μέσα πίεσης, θερμοκρασίας και χρόνου για να εξασφαλίζεται πλήρης αποστήρωση. Δεν ξέρω, αυτή η μέθοδο δεν υπάρχει. Είναι η καλύτερη μέθοδο από ό,τι ξέρω. Εκτό αν μου πει κανεί ότι δεν ισχύει πλέον αυτή η μέθοδο. Είναι μια μέθοδο που ε, φωνεύει οποιαδήποτε πηγή ε, μικροβίων για να αποφεύγουμε τις ε, ζωνόσους. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν καλύτερη υποστήριξη, να έχουμε καλύτερη παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε αυτάρκεια στην παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργιών για να μπορούμε να ταΐσουμε όλα τα ζώα ε, που εκτρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ντάγμα. Ωραία, θα δώσω το λόγο τώρα στην ε, Επιτροπή, στον κύριο Ρικ Βιλέμς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή είναι εξαιρετική και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, το έχουμε πει ήδη σε μια προηγούμενη συνεδρίαση. Να επανέλθω όμως σε κάποια σημεία τα οποία ανέφερε ο εισηγητής στην εισαγωγή του και να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο. Ο εισηγητής πολύ σωστά έθιξε ένα πολύ ε, καλό σημείο. Ιστορικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη εισαγωγή, εισαγωγέας σόγιας και πλακούντων σόγιας. Από το 2009, 2010 η Κίνα μας έχει ξεπεράσει. Επομένως ε, δεν είμαστε ακριβώς το ίδιο σημείο με τους εταίρους μας. Δεν... Ε, η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη εισαγωγέας σόγιας και πλακούντων σόγιας. Άρα εκεί δεν μπορούμε εμείς να, κάνουμε, να παίξουμε παιχνίδι αν θέλετε. Και επίσης προτείνει ο εισηγητής να κάνουμε μία μελέτη για τις ζωικές πρωτεΐνες. Αυτό είναι ένα θέμα ταμπού εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια. Ίσως έπρεπε όμως να το ξανασκεφτούμε γιατί είναι μία, μία αμεληταία πηγή πρωτεϊνών. Άρα θα πρέπει το ελάχιστο που να κάνουμε είναι να αναλύσουμε. Είπατε ότι για λόγους οικονομικούς το να παράγουμε πρωτεΐνες ίσως να μην είναι ιδιαίτερα αποδοτικό όπω όπως με τα δημητριακά. Ίσως να έχετε δίκιο. Όμως για τα πρωτεϊνούχα εδώ και ένα χρόνο οι τα εδάφη, τα καλλιεργούμενα αυξάνονται. Δεν μιλάμε ότι αυξάνονται με μεγάλους ρυθμούς, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια κάποια επιστροφή. Έχουμε το άρθρο 68 του, ε, κανονικού, του οριζόντιου κανονισμού που επιτρέπει να, στα κράτη-μέλη να πάρουν κάποια μέτρα και έχουμε στη Γαλλία και στην Πολωνία μια αύξηση των καλλιεργουμένων εδαφών. Αναφερθήκατε στους ε, γενετικά τροπομενούς οργανισμούς. Όμως εισάγουμε γενετικά τροποποιημένη σόγια που εγκρίνεται, που είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εισάγουμε μία εγκεκριμένη σόγια. Επίσης, ε, και αναφέρατε εσείς και άλλοι συναδελφοί σας, ότι είναι μια συζήτηση που μας απασχολεί εδώ και χρόνια, όχι 13, 20 χρόνια μιλάμε για τις πρωτεΐνες. Και στο παρελθόν είχαμε αναπτύξει διάφορους τρόπους που μας επέτρεπαν να υποστηρίζουμε την παραγωγή πρωτεϊνούχων, είτε όσπρια, πρωτεϊνούχα, ε, ξηρές ζωοτροφές κτλ. Όλα αυτά όμως ήταν μέτρα τα οποία ήταν ιδιαίτερα δαπανηρά και δεν ήταν καθόλου αποδοτικά. Και από την άλλη πλευρά, παρά την ε, ε, και παρόλα αυτά το, η ζήτηση για τη σόγια και για τους πλακούντες σόγιας ε, αυξά, αυξάνεται και θα αυξάνεται όσο αυξάνεται και η γνωτροφία στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια με, το, με τα αιτήματα για βιοεθέρες για την παραγωγή κράμβης, ε, βλέπουμε, και με την παραγωγή κράμβης βλέπουμε ότι καλύπτουμε κατά 30 έως 35% της ανάγκης μας σε πρωτεϊνούχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί λιγάκι τα τελευταία χρόνια, μια και έχουμε μεγαλύτερες ε, εκτάσεις που καλλιεργούνται με κράμβη, λόγω ακριβώς αυτής της ζήτησης για βιοεθέρες, βιοεστέρες. Ε, τώρα, τι μπορούμε, εάν λάβουμε υπόψη μας τη σόγια και τους πλακώντες, τις πλακούντες σόγιας, ε, μπορούμε να βάλουμε μια τάξη, γιατί εισάγουμε 30 με 35 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμο σόγιας ε, κάθε χρόνο. Αυτό το είναι 40 εκατομμύρια τόνοι σόγιας με το ισοδύναμο, αν το αλλάξουμε λαμβάνοντας υπόψη και την απόδοση, μία απόδοση 2,8 ή 3, 3 τόνους ανά εκτάριο, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 14 εκατομμύρια εκτάρια να καλλιεργούνται με σόγια παραπάνω από τη σήμερα για να έχουμε μία κάλυψη. Άρα, αυτά τα 14 εκατομμύρια εκτάρια πού θα τα βρούμε. Καταρχάς θα πρέπει να τα, να τα πάρουμε από τα δημητριακά, τα σιτηρά. Η σίκαλη αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν βλέπω και πολλά εκτάρια να φερόνται στην καλλιεργία της ε, σίκαλης. Για τα το να πάρουμε ε, κάποια εκτάρια. Άρα όμως ε, θα πρέπει να χάσουμε κυρίως μαλακό στάρι. Λαμβάνοντας υπόψη είναι ότι 14 εκατομμύρια εκτάρια είναι το, τα 2 τρίτα των εκτάσεων που καλλιεργούνται με μαλακό στάρι, τι θα κάνουμε, Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει, είναι καθαρή εξαγω, εξαγωγέας 10 εκατομμυρίων τόνων μαλακού σταριού. Οι εισαγωγές μας θα πρέπει να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο με τις εισαγωγές, άρα έχουμε 10 εκατομμύρια τόνους ε, ισοδύναμου, δηλαδή 6 τόνους το εκτάριο, δηλαδή 1,5 εκατομμύρια εκτάρια, που θα πρέπει να τα συγκρίνουμε με τα 14 εκατομμύρια εκτάρια οποίο έχουμε ανάγκη. Άρα πάρα πολύ δύσκολο θεωρώ να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει αυτάρκης στις πρωτεΐνες. Γιατί θα έπρεπε να εισάγει πλέον μαλακό στάρι. Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι μια ρεαλιστική λύση. Όταν συζητήθηκε το θέμα αυτό σε μια προηγούμενη συνεδρίαση, η ανακοίνωση για την κοινή γεωργική πολιτική για το μετά το 2013 δεν είχε ανακοινωθεί, δεν είχε δημοσιευθεί. Να σας, να σας δώσω ένα μήνυμα τώρα. Στην ανακοίνωση αυτή, στο κεφάλαιο που αναφέρεται για την, στην διατροφική ασφάλεια, ένα σημείο λέ, αναφέρεται στις πρωτεΐνες και λέει εκεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις συνεργασίες, τις συνέργειες ανάμεσα στην, ε, στις καλλιέργειες, ε, στην εκτροφή ε, μέσω των πρωτεϊνών. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μια ανάλυση από τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Σας θυμίζω όμως ότι αν θέλουμε να αντεκαταστήσουμε όλες τις εισαγωγές της σόγιας θα πρέπει να αφιερώσουμε 14-15 εκατομμύρια εκτάρια που πρέπει να βρεθούν για να καλλιεργηθεί η σόγια. Άρα θα πρέπει να αντεκαταστήσουμε άλλες καλλιέργειες. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις, λέει η Πρόεδρος, πολύ ενδιαφέρουσας για την συζήτησή μας. Ποιο θέλει να ζητήσει το λόγο. Ε, Το συγγνώμη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο προλαλής σας ε, και η Κομισιόν. Το πρόβλημα είναι να μην χρησιμοποιούμε ε, απόβλητα ζώων για τα μη μυρικαστικά, διότι ούτως ή άλλως χρειάζεται ένα, μια ανάμιξη, ένα μείγμα όλων των. Να χρησιμοποιούμε τώρα μόνο φυτικά, ε, φυτικές πρωτεΐνες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ δεν έχω ξαναδιαβάσει, οφείλω να ομολογήσω όλες τις ε, διατάξεις ε, του 2001, παραδείγματος χάρη, αλλά φαντάζομαι ότι εάν δεν δίνουμε άλευρα ζωικής προέλευσης από ψάρια, από γαρίδες κτλ. στι στις καλλιέργειε δεν θα μπορέσουμε να παράγουμε ψάρια. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Κάτι άλλο το οποίο δεν θεωρώ ότι έχει ζητηθεί επί μακρόν και λεπτομερώς είναι το θέμα της χρησιμοποίησης των αποβλήτων ζωικής προέλευσης. Ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εδώ. Για το, στο κείμενο αυτό εδώ θέλουμε να καλέσουμε, ε, να ζητήσουμε μάλλον την χρήση των ε, ζωικών αποβλήτων για το, ε, για το αέριο, ε, για το βιοαέριο όμως ταυτόχρονα μιλάμε και για το διοξίδιο του άνθρακα. Δηλαδή ναι μεν λέμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερο βιοαέριο αλλά βάζουμε διαφορά αν είναι ζωικής προέλευσης ή φυτικής προέλευσης ε, ε, η πρώτη, το, η πρώτη ύλη, τα απόβλητα δηλαδή. Και εάν χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα απόβλητα, ναι με να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να, χρησιμοποιήσουμε τα απόβλητα αυτά για να παράγουμε βιοαέριο, παράγουμε όμως ταυτόχρονα, δηλαδή να παράγουμε ενέργεια, παράγουμε όμως ταυτόχρονα και τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια γραμμή θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτού του είδους ενέργειες τις ε, υποστηρίζουμε ή όχι ε, και μέχρι ποιο βαθμό τις υποστηρίζουμε διότι τα απόβλητα αυτή τη στιγμή τα χρησιμοποιούμε ε, συγγνώμη, ναι, τα αυτά τα απόβλητα μαζί με την παραγωγή ολοκλήρων περιοχών ας πούμε με σιτηρά για να παράγουμε βιοαέριο. Απ' την άλλη πλευρά όμως τι κάνουμε με το διοξείδιο του άνθρωπου το οποίο εκλείεται. Μπορούμε να το συλλέξουμε ή όχι. Η Κατρίν Σουγέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ζήτημα αυτό των πρωτενών είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις εισαγωγές ε, σόγιας, πλακούντας σόγιας και άλλων πρωτεϊνούχων, διότι βάζουμε σε κίνδυνο την διατροφική μας ασφάλεια και εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο για την ε, διατροφή μας από εκτός Ευρώπης χώρες. Έχω να κάνω μια παρατήρηση προς τον εισηγητή, τον κύριο Ταβάτζη. Αναρωτιέμαι, πρέπει να επενθυμίζουμε στο κείμενο αυτό το τραγικό, την τραγική εκείνη περίοδο της και φελοπάθειας των βοηδών. Γιατί να τα βάζουμε με τα ζώα και με μια κατηγορία ζώων που κατά τα άλλα μας δίνουν εξαίρετα προϊόντα. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει διατροφική ασφάλεια από το κρέας, να προωθήσουμε τις φυτικές πρωτεΐνες, ναι, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αποφύγουμε τις ζωικές πρωτεΐνες. Κάτι για το οποίο στηρίζω τον εισηγητή είναι ότι δεδομένων των ποσοστώσεων εισαγωγών πρωτεϊνούχων και κυρίως σόγιας πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά την προέλευση των πρωτεϊνούχων ουσιών που εισάγονται στην Ευρώπη. Να ενισχύσουμε τις επιθεωρήσεις επίσης επιτόπου. Γιατί λοιπόν η παράγραφος 4 είναι διατυπωμένη έτσι χλιαρά όπου λέμε ότι ο μηχανισμός ελέγχου της προέλευσης των πρωτεϊνούχων καλλιερών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που λέει εδώ ότι δίνει ένα δυνητικό όρο, ενώ πρέπει να φαίνεται ότι συστηματικά ζητάμε να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και όχι μερικές φορές μόνο. Ο συγκεκριτής μας, ο κύριος Σταβάτζη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά σχετικά με τον προβληματισμό σας. Πιστεύω ότι πρέπει να επιστήσουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας στο θέμα της αλλαγής στην οτροπία διατροφής των Ευρωπαίων πολιτών. Είτε πρόκειται για την παχυσαρκή, είτε πρόκειται για άλλα προβλήματα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έπειτα, για την διατροφική ασφάλεια, μια που είμαστε ευάλωτοι και εξαρτόμεστα από εξωτερικές αγορές, συμφωνώ επίσης απόλυτα μαζί σα και με του άλλου συναδέρφους. Σε αυτά που είπε η Ντάκμα Ροτμπέρεντ, θέλω να τη ζητήσω να στηρίξει την τροπολογία που θα υποβάλω στην έκθεση αυτή. Γιατί βλέπετε είμαι πλήρε μέλο στην Επιτροπή Γεωργίας και σκιώδης εισηγητή στην Επιτροπή Γεωργίας, αλλά εισηγητή για γνωμοδότηση εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Υποβάλλω λοιπόν τροπολογία με την οποία προτείνω να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει, να εκπονήσει μελέτη για το θέμα των ζωικών αποβλήτων όσον αφορά τα μη μυρικαστικά. Και συμφωνώ επίσης και με την Κατρίν Σουγέ για το ότι δεν πρέπει να αποκλείσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ηχθιάλευρα ή ε, απόβλητα ζωικά για τα μη μυρικαστικά. Γιατί για τα μυρικαστικά το έχουμε αποκλείσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τα ζώα που δεν είναι μυρικαστικά όμως, πρέπει να το δούμε. Δεν είναι δυνατόν να εξακολουθούμε να ζούμε με τέτοια ταμπού. Για τον κύριο Ρώση. Ήμουν εισηγητής για το βιοαέριο και συμφωνώ με την Τάγμαρ. Είναι αλήθεια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τις ζωικές πρωτεΐνες και για το βιοαέριο. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά αλλά είναι πολυτέλεια να μην χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα ζωικά απόβλητα για τις ζωικές πρωτεΐνες. Εδώ υπάρχει συνένεση για το ότι, και το είπε και εκπρόσωπος της Επιτροπής, για το ότι ποτέ δεν θα έχουμε αρκετή παραγωγή πρωτεϊνών στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο. Και είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε όρια 40 εκατομμύρια εκτάρια για τις φυτικές πρωτεΐνες. Γι' αυτό πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα στις ζωικές πρωτεΐνες για τα μη μυρικαστικά. Σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι και στην Επιτροπή Γεωργίας θα έχουμε μία μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση απέναντι στις ζωικές πρωτεΐνες, περισσότερη ακόμα από ό,τι εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Γι' αυτό ήθελα να είμαι προσεκτικός ε, στη διατύπωση της γνωμοδότησής μου, γιατί πίστευα ότι υπήρξε μεγάλη αντίσταση από πλευρά σας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής όμως που διαπιστώνω ότι είσαστε πιο ρεαλιστές και υιοθετείτε μια πολύ πραγματιστική θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά για την ποιότητα της έκθεσής σας και ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή σας στην ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Η προθεσμία είναι 7 Δεκεμβρίου. 25 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε εδώ, στη Γεωργία 26 και 27 Ιανουαρίου και στην Ολομέλεια θα πάει η έκθεση αυτή τον Μάρτιο του 2011. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι προγράμματα πολιτικής συνοχής 2007-2013. Ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά, αν μου επιτρέπετε. Στην συνθήκη της ε, Λισαβόνας καθορίζεται μια βασική αρχή που είναι η προώθηση της ε, εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Αυτό λέει το άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Έχει περάσει ένα χρόνος ήδη από την στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας. Και να δούμε τι γίνεται με την πολιτική συνοχή, με τις πολιτικές γιατί ούτως ή άλλως όλα αυτά συνδέονται με την ε, οικονομική, κοινωνική ε, και οικονομική συνοχή. Διότι υπάρχει και μια περιβαλλοντική επίσης πτυχή. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ε, υπογραμμίσουμε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή των πολιτικών συνοχής είναι τελείως απαράδεκτη, διότι ε, έχουμε μονάχα το 21% του συνόλου των επιλεγέντων προγραμμάτων έχει εφαρμοστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με τη στρατηγική του 2020, κυρίως ε, προγράμματα που αφορούν τον περιορισμό της ε, εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα ή την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. όλα αυτά τα, όλα αυτά τα προγράμματα που αφορούν ε, στην ε, στρατηγική 2020 είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα παρακολουθήσουμε από κοντά. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι ένα θέμα καυτό θα έλεγα. Ακούστηκε ένα ποσοστό 30% μείωση. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος έχει ε, δημοσιευθεί. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη μας, είναι ζωτική σημασίας να αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα όσο να το νωρίτερα και θα πρέπει να επιταχύνουμε και τους ρυθμούς ε, εφαρμογής. Ένας άλλος στόχος είναι η προώθηση πράσινων θέσεων απασχόλησης θα πρέπει μέσω αυτών των προγραμμάτων να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και ούτως ή άλλως αυτές οι θέσεις απασχόλησης αφορούν ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής ε, του 2020. Επίσης θα πρέπει να να προωθηθούν προγράμματα που να συμβάλλουν στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών ή ε, τομέα, τομέας πρόληψης και της αποκατάστασης βιομηχανικών ζωνών. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια επιτάχυνση αν θέλετε, διότι έχουμε χαμηλό βαθμό εφαρμογής και υλοποίησης των προγραμμάτων. Αυτό επίσης το ε, οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει την ευκαμψία των κανόνων που αφορούν την εκτέλεση των προγραμμάτων γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μειωθεί και είναι εφικτό να μειωθεί η γραφειοκρατία. Προφανώς όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα πλαίσια των κανόνων και της ισχύουσας νομοθεσίας. Όμως θα πρέπει να προωθήσουμε, αν θέλετε, την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η διαφάνεια και κυρίως στον περιβαλλοντικό τομέα πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα, ποια είναι τα project τα οποία υιοθετήθηκαν και τι έχει εφαρμοστεί από όλα αυτά. και να το δούμε και με θετικό, από, από την θετική πλευρά και από την αρνητική. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε καταρχάς ποια είναι τα project τα οποία έχουν ε, υιοθετηθεί και να δούμε ποια από αυτά έρχονται σε αντίθεση με τους ε, στόχους που έχουμε θέσει για την ενέργεια ή για το περιβάλλον. Δηλαδή, εναντίον των στόχων που έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα project τα οποία έχουν υιοθετηθεί και τα οποία υπηρετούν τους στόχους του 2020. Άρα, τα project θα τα δούμε και από τις δύο πλευρές και αυτά από την, να δούμε τα project τα οποία έρχονται σε αντίθεση ε, με τους στόχους μας και αυτά που συνδράμουν το έργο μας. Διότι ο ελάχιστο κοινό παρονομαστή, μάλλον το στοιχείο το οποίο μα ενώνει όλου, είναι η στόχοι τη στρατηγική για το 2020. και θα πρέπει δηλαδή να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση, ε, να δούμε ποια είναι τα project τα οποία έχουν υιοθετηθεί και ποια έχουν εφαρμοστεί. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα project τα οποία έχουν εγκριθεί και ποια από αυτά που έχουν εγκριθεί έχουν ε, υλοποιηθεί, έχουν εφαρμοστεί. Με τον τρόπο αυτό προωθούμε και την διαφάνεια αλλά και την σωστή επίβλεψη, τον σωστό έλεγχο. Θα ήθελα να ήθελα, να να ευχαριστήσω και τον ε, σκιώδη εισηγητή, τον κύριο Μίκο Λάσιτς, με τον οποίο ε, έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά. γιατί πραγματικά συνεργαζόμαστε για να υποβάλουμε την καλύτερη δυνατή έκθεση για ένα θέμα που είναι τόσο σημαντικό και στο οποίο αφιερώνεται το 1 τρίτο της κοινοτικής χρηματοδότησης. Η κυρία Σίλντερς, λέει πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότηση που μα έχει παρουσιάσει. Η πολιτική συνοχή είναι μία από τι πιο επιτυχημένε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα από του λόγου για του οποίου η διεύρυνση του 2004 ήταν τόσο επιτυχή. και από την ε, δική μου εκλογική περιφέρεια στην Ιρλανδία διαπιστώνουμε πόσο επιτυχημένη είναι και πόσο μα έχει βοηθήσει η πολιτική τη συνοχή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ανισότητε που δεν έχουν εκλείψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν θέματα μη βιώσιμη ανάπτυξη και ανεπάρκεια. Τώρα για την εφαρμογή των προγραμμάτων από το 2007 μέχρι το 2013 σε αυτήν την περίοδο προγραμματική περίοδο, εξετάζουμε τρόπου για να έχουμε καλύτερα και πιο, καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή στον περιβαλλοντικό τομέα και χαιρετίζω το ότι ο εισηγητή το έχει αναφέρει αυτό το σημείο στην έκθεσή του. Θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ιδίω σε αυτή την περίοδο κρίση που πιέζει τι εθνικέ κυβερνήσει. Ο εισηγητή θα πρέπει να προσπαθήσει η κοινή γνώμη να στραφεί ε, στην ε, έλλειψη προγραμμάτων συνοχή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα έχω κατά νου ε, τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Θέλουμε, όπως περιγράφεται στην Στρατηγική Ευρώπη 2020, να, έχουμε, να καταργηθούν όλες αυτές οι ανισότητες. Οι πολιτικές συνοχής είναι άλλο ένα αυτό παράδειγμα του τι διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια απλή Ένωση Χωρών για Εμπορικού Στόχου όπω είναι αυτά. Πρέπει να προσπαθήσουμε τι επιτυχίε που έχουμε επιτύχει να τι επεκτείνουμε και μετά το 2014. Για άλλη μια φορά, συγχαίρω τον εισηγητή για το έγγραφο αυτό και περιμένω να εργαστώ με του συναδέλφου μου για το έγγραφο αυτό τι επόμενε εβδομάδε. Ρίχαρτ Ζέμπερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο για την έκθεση και νομίζω ότι πρέπει στην περιφερειακή πολιτική και στην πολιτική συνοχή να φροντίσουμε να υπάρχει ενιαίο πνεύμα και να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση και ενερμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής 2020. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό και θα είναι και στο μέλλον πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου όλα τα έργα και όλα τα προγράμματα να είναι ε, κατευθυνόμενα προς αυτό το στόχο. Και ε, αυτό θα είναι και ένας στόχος για την επόμενη προγραμματική περίοδο και θα μας απασχολήσει όταν θα πρέπει να δούμε πόσα χρήματα θα χρειαστούμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την υλοποίηση κατά την τρέχουσα περίοδο. Και γι' αυτό ε, ένα σημείο που είναι ενδιαφέρον είναι η απλούστευση των πόρων, ε, η απλούστευση των διαδικασιών για τη χορηγήση των πόρων. Αγαπητοί συνάδελφοι, Λίγο ησυχία παρακαλώ για να μπορέσει ο συνάδελφος. Ε, οι πράσινοι έχουν πάντοτε σημαντικέ συζητήσεις και δεν έχουν χρόνο να ακούσουν εμένα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μιλάμε εμείς. Η περιφερειακή πολιτική μάλλον δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πρασίνους. Τέλος πάντων, αστιαύομαι, αστιαύομαι, συγγνώμη. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα που συζητούσαμε. Είναι σημαντικό για μας να έχουμε ε, μια περιφερειακή προσέγγιση και οι περιφέρειες γνωρίζουν καλύτερα οι ίδιες πώς θέλουν να διαμορφώσουν ε, τις τοπικές τους κοινότητες και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Στρατηγική θα πρέπει να έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να το καταφέρει. Αυτή η χρηματοδότηση βέβαια για να ξεκινήσει η ανάπτυξη πρέπει να είναι χρηματοδότηση για να ξεκινήσει μόνο και μετά θα πρέπει να είναι βιώσιμα τα προγράμματα μακροπρόθεσμα από μόνο και αυτό νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε ώστε ε, ε, να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και με, το, τα θέματα ε, των ε, πυρκαγιών στα δάση και των φυσικών καταστροφών είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα ε, τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια βιώσιμη πολιτική που θα εκμεταλλεύεται σωστά του πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες γιατί εδώ έχουμε αρμοδιότητα των κρατών μελών που πρέπει να φροντίσουν για τα προβλήματα αυτά και νομίζω ότι δεν θα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει το πλήρες καθήκον σε αυτό το θέμα. πολύ συχνά υπάρχουν απλές εθνικές νομοθεσίες ή απλοί κανονισμοί που θα μπορούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα πολύ απλούστερα. Το να μην ε, υπάρχει ε, δυνατότητα να χτίσει κανείς σε περιοχές όπου έχουν υπάρξει πυρκαγιές για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτό είναι μια σωστή διάταξη που πιστεύω ότι θα δώσει καλύτερη απόδοση και στα χρήματα που θα πανάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική μας έχει βοηθήσει να έχουμε καλύτερες υποδομές, να έχουμε ε, καλύτερη περιβαλλοντική προστασία και αυτό είναι ένας ιδιαίτερος στόχος για τη δική μας Επιτροπή. Όπως ε, είπαμε όμως και πάλι, τα κράτη-μέλη που επωφελούνται από την, από την πολιτική αυτή θα πρέπει στις δικές τους νομοθεσίες να μην ξεχνούν αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ. Ε, Ένα λόγος είναι ότι, ε, και απαντώ έμασα και στον συνάδελφο πριν που έκανε τα σχόλια για τους πράσινους, ότι οι πράσινοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την ε, περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχής και μάλιστα γνωρίζω και στον συνάδελφο ότι είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης η οποία δυστυχώς, και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, να πω ότι συνεχώς και από την πρώτη στιγμή γίνεται ακριβώς τις ίδιες ώρες με την Επιτροπή ε, για το Περιβάλλον, ε, στην οποία συζητάμε επίσης ενδιαφέροντα ζητήματα και δεν μπορώ να τα αποκριθώ και στις δύο. Αυτή τη στιγμή εγκατέλειψα ε, την ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που μιλάμε για την πολιτική συνοχή, τον υπολογισμό, τις συνέργειες, τις νέες πρωτοβουλίες για να ακούσω ακριβώς αυτά που λέγονται σε αυτή την ε, Επιτροπή σήμερα προφανώς και υπερασπίζουμε την ε, ε, πολιτική συνοχής, μόνο που σήμερα στην εποχή της ε, οικονομικής κρίσης χρειάζεται μια γενναία ανασύνταξη και ακριβώς γιατί η κρίση είναι και οικονομική που τη βλέπουμε σαν ντόμινο να εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τουλάχιστον τον Ευρωπαϊκό Νότο αλλά ταυτόχρονα εκτός από η οικονομική κρίση αυτή είναι και περιβαλλοντική και ενεργειακή και κοινωνική. Άρα χρειάζεται συνολικά αλλαγή πολιτικών και δεν μπορούμε να τις έχουμε με τις συγκεκριμένες πολιτικές της σοσιαλφιλελεύθερης συνένεσης που διαβλέπουμε και στην πολιτική της ε, Επιτροπής Μπαρόζο. Υπάρχουν λοιπόν ανάγκη για συνέργειες, για αυξημένη αποτελεσματικότητα ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, άλλων διαρθρωτικών ταμείων, υπάρχουν ανάγκη, υπάρχει ανάγκη για αναθεωρήσεις στην πολιτική και προφανώς το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας και ε, το οποίο αποτελεί απλώς και κάποιες πρώτες σκέψεις, ένα σκελετό ε, και έτσι τον εμείς το αντιμετωπίζουμε. Το κείμενο δηλαδή το, που είναι και η αφορμή της σημερινή συζήτηση θέλει έναν γενναίο εμπλουτισμό και θα καταθέσουμε τροπολογίες προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Θέλουμε να δώσουμε αυτή την άλλη προοπτική στην ε, πολιτική συνοχής και να αμυνθούμε απέναντι σε αυτές τις αντιλήψεις που μιλούν από διάφορους κύκλους συμφερόντων ή και από χώρε για επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής. Υπάρχει, υπάρχει ανάγκη να ε, εμβαθύνουμε και να δώσουμε ε, βάρος και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα τοπικά, τα περιφερειακά, τα εθνικά που υπάρχουν. Υπάρχει ανάγκη να συνδέσουμε και θα το ακούσετε φυσικά αυτό και από εμά και από την Επιτροπή εδώ που υπάρχει η ευαισθησία να υποστηριχθεί ο στόχος του 30% μείωση ε, για, τον, για να ανταποκριθούμε στις ε, προοπτικές και στο πρόβλημα της ε, κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει ανάγκη να συνταυτίσουμε, να συμπεριλάβουμε τους στόχους για την προστασία τις βιοπικιλότητες. Και όπως ε, ξέρουμε η χρονιά αυτή που τελειώνει ήταν αφιερωμένη στο θέμα αυτό. Υπάρχει ανάγκη να περάσουμε σε δείκτες και σε πολιτικές πέρα από τα φτωχά μέτρα του GDP. Δηλαδή υπάρχουν άλλα ζητήματα που πρέπει να εμπλουτίσουν τις, ε, α, ε, τις προσεγγίσεις μας ακριβώς γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε ένα τροχαίο ατύχημα μπορεί να αυξήσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Ακριβώς γιατί θα δουλέψουν τα νοσοκομεία, θα δουλέψουν τα γραφεία κηδιών και στο τέλος αν κόψουμε όλα τα δάση της Ευρώπης και τα κάνουμε χαρτί ή τα πουλήσουμε στο εξωτερικό, αυτοί οι δείκτες θα ανέβουν. Η ίδια η ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, το μέλλον του πλανήτη θα υποβαθμιστεί. Χρειάζεται λοιπόν νέες προσεγγίσεις που να βάζουν και τον άνθρωπο στο επίκεντρο, αλλά και το περιβάλλον και το μέλλον του πλανήτη. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό στη συνέχεια και στην Επιτροπή μας και με αφορμή το θέμα που συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μύροσλαφ Μικολάσιτζο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο, διότι όπως είπε και όπως και ο αγαπητός μου συνάδελφος κύριος Τρεμόπουλος είμαστε και στις δύο επιτροπές και στην περιφερειακή και εδώ και εγώ το ίδιο ε, και, εμένα, και με μένα το ίδιο συμβαίνει θα ήθελα να πω αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον Χωζέ Μανουέλ Φερνάντες, ε, ότι με έναν πάρα πολύ εύπεπτο και ξαφή τρόπο μας ενημέρωσε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές σε αυτή την έκθεση, την έκθεση που είμαι ο βασικός, ε, γιατί είμαστε, είμαι εισηγητής επί της ουσίας εγώ. Επειδή είμαι ένα πληρωματικό μέλος αυτής της Επιτροπής και κύριο μέλος ε, της Επιτροπής Περιφερει... της Περιφερειακής Πολιτικής, ε, θα σας, υπόσχομαι ότι θα συμπεριλάβω όλα όσα ακούστηκαν εδώ στην τελική εκδοχή της έκθεσης. Δηλαδή θα υπάρχει και η συνιστόσα της, ε, περιβαλλοντικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η έκθεση αυτή δείχνει ακριβώς πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πολιτική για τη συνοχή. Εμείς προσπαθούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να δούμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η πολιτική στο μέλλον. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προχωρούμε, προχωρούν οι εργασίες ε, ε, σε αυτή την έκθεση ήρθα, έχω έρθει σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, ο κύριος Νόπουλος δεν ήταν παρόν, αλλά ελπίζω θα μου δώσει τη συνειφορά του να τον πιο γρήγορα, έτσι ώστε, όπως υποσχέθηκα νωρίτερα, να μπορέσω να εντάξω τις, όλες τις απόψεις ε, στην έκθεσή μου. στο σχέδιο τουλάχιστον της έκθεσης πριν καταλήξουμε στο, στην τελική έκθεση 11 Ιανουαρίου. Πάντως ε, αυτά τα οποία άκουσα εδώ είναι μια πολύτιμη συνεισφορά για, την για τον περαιτέρω εμπλουτισμό του κειμένου μου και ελπίζω ότι τα αιτήματα τα οποία ε, παρουσίασε ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες στην αρχή ε, αποτελούν και δικές μου προτεραιότητες. Και να ξέρετε ότι αυτές οι προτεραιότητες θα εκφραστούν με πολύ πιο έντονο τρόπο στο κείμενό μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε το λόγο, γιατί με ακούσατε και περιμένω ε, με ιδιαίτερη ανυπομονησία την συνεργασία με όλους και περιμένω επίσης και τις ε, τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ο κύριος... Από πλευρά της Επιτροπής, ο κύριος Πόσο, παρακαλώ. Αλλά σύντομα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω το έργο του εισηγητού και σας ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση εδώ στην Επιτροπή σας. Ο σκοπός ε, αυτής της υποβολής εκθέσεως στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού ήταν το να έχουμε μια στρατηγική και πλήρη συζήτηση της ε, προόδου κατά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις απόψεις που εκφράστηκαν στην Επιτροπή σχετικά με την συμβολή της πολιτικής συνοχής στους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν αναλύουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, Υπολογίζουμε ότι πάνω από 30% των πόρων στην πολιτική συνοχής ε, δόθηκαν σε άμεσες ε, ή έμεσες περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Οι άμεσες περιβαλλοντικές προτεραιότητες είναι αυτές ε, που υπάρχουν στον τομέα του πόσιμου ύδατος, ε, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, αποχέτευσης κλπ. Και οι έμεσες είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οικολογική αποτελεσματικότητα και βιώσιμες πολιτικές μεταφορών συμπεριλαμβανομένης και των καθαρών αστικών μεταφορών. Τα προγράμματα αυτά αυτά ε, γίνονται σε επιμερισμένη διαχείριση και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της αρχής της επικουρικότητας είναι η πολιτική συνοχή. Η στρατηγική λοιπόν έκθεση σχεδιάστηκε ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν εκθέσεις για το πολύ σημαντικό τους ρόλο κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό συνιστώ προς τους ε, κυρίους και κυρίες βουλευτές τις εθνικές εκθέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες ε, στην γλώσσα γλώσσα όλων των κρατών μελών στην ιστοσελίδα μας, γιατί θα έχετε μια πληρέστερη εικόνα των εθνικών δραστηριοτήτων. Αυτή η έκθεση λοιπόν παίζει το σημαντικό ρόλο της διαφάνειας. Όπως βλέπετε από τη στρατηγική μας έκθεση, η Επιτροπή συμμερίζεται ε, τις ανησυχίες για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων, όπου η πρόοδος είναι πιο αργή από ό,τι θα επιθυμούσαμε και ο εισηγητής στην έκθεσή του το τονίζει αυτό. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις διαχειριστικές αρχές ε, για να δημιουργήσει ε, επιτόπου ικανότητες. Συνεργάζεται με την πρωτοβουλία Jaspers για περιβαλλοντικά προγράμματα και επίσης άμεσα συνεργάζεται η Επιτροπή, πολλές υπηρεσίες της Επιτροπής σε δραστηριότητες δικτύωσης με διασκέψεις, σεμινάρια για την βελτίωση των πόρων επιτόπου και προσπαθούμε μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια να ε, συνεργαστούμε για την τεχνική βοήθεια ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις διαχειριστικές αρχές να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι σημαντικό αυτό που αναφέρει ο εισηγητή για, για τις ανάγκες αναπρογραμματισμού και ε, αναλλαγή της συγχρηματοδότηση. Θα φροντίσουμε οι πληροφορίε αυτέ να είναι διαθέσιμε με τρόπο εύληπτο, με χάρτες και γραφικές παραστάσεις και η αποτύπωση με χάρτες της χρηματοδότησης είναι ε, ιδιαίτερα ε, καλή ιδέα και στους επόμενους μήνες που θα επανέλθουμε στην Επιτροπή σας θα έχουμε και κάποια έκθεση πρόοδου για το πώς οι πληροφορίες μπορούν να είναι καλύτερα προσβάσιμες από τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών είναι 9 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ότι η ψηφοφορία εδώ θα γίνει 20 και 25 Νοεμβρίου 2011. Α, ο κύριος Φερνάντες όμως, συγγνώμη κύριε Σιγητά που δεν σας έδωσα το λόγο πριν, βιάστηκα. Κι εγώ θα είμαι σύντομος κυρία Πρόεδρε, μην ανησυχείτε. Σχετικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τόσο είπατε. Ευχαριστώ επίσης και το συντάκτη γνωμοδότησης για το ανοιχτό πνεύμα που επιδεικνύει. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να καταλήξουμε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μιλάμε για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές ετοιμάζεται έκθεση άλλη από την ΕΝΒΗ. Τώρα δεν θα αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν θα μιλήσουμε για αλλαγέ όσον αφορά το έπος κριτήριο για τη χρηματοδότηση κτλ. Μιλάμε για τα ήδη τα κριτήρια. Πάνω σε αυτά δουλεύουμε, με αυτά. στα υπάρχοντα βασιζόμαστε. Το κείμενο λοιπόν εκφράζει την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της στρατηγικής της για το 2020 με συγκεκριμένες δράσεις για την αηφόρο ανάπτυξη πάνω απ' όλα. Υπάρχει φιλοδοξία που συνδέεται με αυτό και που είναι να επιταχύνουμε τη διάθεση των υπαρχόντων κονδυλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάποια ελαστικότητα. Ελπίζω να μην χάσουμε ούτε δεκάρα. Να μπορέσουν όλες οι χώρες να υποφεληθούν μέχρι την τελευταία δεκάρα για προγράμματα που είναι πολύ σημαντικά για την επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας και για τα όσα είπατε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Συνεπώς, έλεγα 9 Δεκεμβρίου υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ψηφίσουμε 24-26 Ιανουαρίου 2011, 20 ε, Φεβρουαρίου στη Ρέγγι και τον Απρίλιο θα πάει στην Ολομέλεια. Ερχόμαστε τώρα στην προφορική ερώτηση της κυρίας Χάση όσον αφορά την καταστροφή από την Ερυθρά Υλή στην Ουγγαρία. Εδώ τίθεται το θέμα εφαρμογή κοινοτικού δικαίου. Ένα τέταρτο θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα για την Αιλή, γιατί έχουμε μετά κι άλλα για την κοινοτική νομοθεσία. Μπλάνκο, Διευθυντή τη Γενική διεύθυνση ΕΝΒΗ και συγκεκριμένα σε σχέση με τη βιομηχανία. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Η κυρία Μπλάνκο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας τα συλληπιτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη θλίψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταστροφή αυτή και την απώλεια ανθρώπινων ζών. Ξέρουμε ότι η Υπουργική Κυβέρνηση έκανε μεγάλες προσπάθειες μετά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε καλύτερα την Ουγγαρία. Με το κέντρο πληροφόρησης, το ΜΙΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκόλυνε την ε, μεταφορά της αλληλεγγύης στα πλαίσια ε, του μηχανισμού αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ομάδα με πέντε εμπειρογνώμονες χρησιμοποιήθηκε επί μία ολόκληρη εβδομάδα επιτόπου για να βοηθήσει. Όσον αφορά τώρα την ομοθεσία που εφαρμόζεται σε τέτοιες εγκαταστάσεις, έχουμε να κάνουμε με τον έλεγχο και την πρόληψη, το MBC, έχουμε να κάνουμε την οδηγία για την διαχείριση εξορρυκτικής ε, βιομηχανίας, έχουμε να κάνουμε με τον κατάλογο των ε, αποβλήτων επίσης και την πρόληψη και τον έλεγχο της ρήπανσης. Η Επιτροπή έστειλε στις 22 Οκτωβρίου επιστολή, δηλαδή μόλις ε, πέρασε το πρώτο στάδιο ανταπόκριση στην κρίση, και γράψαμε στις Ουγγρικές Αρχές προκειμένου να μας στείλουν πληροφορίες για το πώς εφαρμόστηκε η νοτική νομοθεσία εκεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς εφαρμόστηκαν. Η απάντηση στην επιστολή αυτή, υπό την μορφή εκτεταμένης και λεπτομερής επιστολής περιλάβανε πάρα πολλές ε, πληροφορίες, μας έφτασε στις 24 Νοεμβρίου. Σας είπα ότι περιλάμβανε πάρα πολλές πληροφορίες, τεχνικές και άλλες και εξακολουθούμε να είμαστε στο στάδιο αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών που μας στείλανε. Εισαγωγικά λοιπόν κυρία Πρόεδρε, Θέλω να σταθώ σε αυτό μόνο και από εκεί και πέρα να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχουν οι εξώτιμοι ευρωβουλευτές. Να τελειώσω υπογραμμίζοντας πάντως την ανάγκη που υπάρχει για μια ορθή και πλήρη εφαρμογή των διαφόρων οδηγιών γενικά της κοινοτικής νομοθεσίας όταν πρόκειται για προστασία από τέτοια ατυχήματα και συμβάντα, έτσι ώστε τέτοιου είδους ατυχήματα να μην επαναληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ταμπάτζη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και έχει να κάνει με την επικινδυνότητα της ερυθράς ηλίας. Πρέπει να θυμίσω στην Επιτροπή ότι υπάρχει συμφωνία της Βασιλείας, η οποία λέει ότι στην περίπτωση όπου υπάρχουν 11,6% pH ε, ή πιο ψηλό ακόμα, τότε θεωρείται επικίνδυνη η ύλη αυτή. Η ρύθμιση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία αυτή της Βασιλείας. Δεύτερον, την προηγούμενη φορά το συζητήσαμε ήδη ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια υποχρεωτική ασφάλιση. Διότι βλέπετε το εργοστάσιο αυτό είναι αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι της τάξης των 42 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε ποια είναι η αναλογία. Ακόμα δηλαδή και αν πουλούσαμε ολόκληρο το εργοστάσιο δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε το κόστος από τη ζημιά που έχει προκληθεί. Υπάρχουν και στα Δυτικά Βαλκάνια και αλλού τέτοιου είδους εργοστάσια. Βοξίτη, εργοστάσια Βοξίτη για παράδειγμα. και το περιβάλλον ξέρουμε ότι έχει την ίδια σημασία όπου και αν βρίσκεται στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό της ερυθράς ηλίας λοιπόν είναι ένα περίπλοκο θέμα και γι' αυτό και εγώ υπέβαλα γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω επιτέλους να μου δώσουν μια απάντηση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μπαρτ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Επιτροπής, όμως η κυρία Χασισάτο δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε την αντικαθιστώ εγώ. Εκείνη υπέβαλε την προφορική ερώτηση. Και τελικά δεν έχουμε ακούσει εδώ καμία συγκεκριμένη απάντηση στις συγκεκριμένες ερωτήσεις της κυρίας Χάση. Υπάρχουν τέσσερις νομοθεσίες, οδηγίες. Εφαρμόζονται εντάξει, 28 Οκτωβρίου στείλατε επιστολή, τέλη Νοεμβρίου πήρατε απάντηση από ό,τι μας είπατε, αλλά οι συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Επίτροπη είναι πρώτα απ' όλα. Μπορούμε γρήγορα να έχουμε μια αξιολόγηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιστολή που πήραν από την Ουγγαρία, για να ξέρουμε τι βήματα πρέπει να αναλάβει το Κοινοβούλιο μας στη συνέχεια. Έπειτα στις συγκεκριμένες ερωτήσεις της κυρίας Χάση είναι ότι η Επιτροπή είναι διατεθειμένη ναι ή όχι να συγκροτήσει ομάδα εργασίας ε, και να την στείλει επιτόπου για να εκτιμήσει την καταστροφή στην Ουγγαρία. Γιατί δεν το κάνει. Άλλη ερώτηση που δεν απαντήσατε είναι όσον αφορά ποια είναι η κατάσταση σε άλλες χώρες. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και αλλού ε, τέτοιες εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες Καπονιά. Η ερώτηση λοιπόν είναι, υπάρχει απογραφή της κατάστασης, ποιες είναι αυτές οι χώρες στην Ευρώπη και υπάρχει διαθέσιμη για το κοινό. Υπάρχουν δηλαδή τοποθεσίες στην Ευρώπη όπου κινδυνεύουμε να έχουμε ένα αντίστοιχο ατύχημα. Μια άλλη ερώτηση της κυρίας Χάση και πολύ σωστά είναι να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή κοινοτικών επιθεωρήσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει και τον Νοέμβριο του 2008 εδώ. Και ψήφισμα είχαμε κάνει και στο άρθρο 4 του ψηφίσματος αυτού, ως Κοινοβούλιο, ως Ολομέλεια, είχαμε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία νομοθετική πρόταση, μια οδηγία για να έχουμε πιο συστηματικά διεξαγωγή κοινοτικών επιθεωρήσεων. Έχουμε φτάσει τέλη 2010. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου, θα φροντίσει να υπάρξει το νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή κοινοτικών επιθεωρήσεων και τι μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσατε, οριζόντιες οδηγίες, κάτι άλλο, ειδική νομοθεσία. Αυτή είναι επίσης λοιπόν μια συγκεκριμένη ερώτηση στην οποία δεν ακούσαμε απάντηση. Επίσης, όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές ασφαλίσεις, ούτε εδώ πήραμε καμία απάντηση. Μπορούμε να περιμένουμε μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Τέλος, η οδηγία με τον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων. Σε μια προηγούμενη συζήτηση είπαμε ότι ο κατάλογος αυτός ακολουθεί κάποια κριτήρια. Μεταξύ άλλων, ως κριτήριο είναι οι επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται. Όμως δεν φτάνει αυτό. Είχαμε πει ότι πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες εφόσον έχουν πάνω από 1% διαβρωτικές ουσίες μέσα. Το του αζότου, για παράδειγμα, που έχει διαβρωτικές ιδιότητες. Μπορεί λοιπόν να μας επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ύλη στην Ουγγαρία μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο απόβλητο. Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις μας γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα το γύρμα. Σε ευχαριστούμε πολύ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και εγώ ζητάω να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, παρακαλώ, στις συγκεκριμένες μας ερωτήσεις. Θα σας ξαναδώσω το λόγο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είσαστε σε θέση να μας απαντήσετε σήμερα, αλλά να ορίσουμε μια άλλη ημερομηνία όπου θα έρθετε και όπου συγκεκριμένα θα μας απαντήσετε. Παρακαλώ, κυρία Μοσετή τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο πλαίσιο όλων αυτών των καταστροφών που έχουν προκληθεί από αμέλεια σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, θα ήθελα να θίξω το θέμα της ε, λήψης μέτρων για την επανόρθωση. Τι μηχανισμός υπάρχει και πώς εφαρμόζεται. Υπάρχει ο μηχανισμός αλληλεγγύης που μπορούμε να κινήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση είναι τεράστια η φυσική καταστροφή και έχει προκληθεί ζημιά όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και στο περιβάλλον. Ισχύει συνήθως η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Από όσο γνωρίζω και ίσως οι συνάδελφοι από την Ουγγαρία μου πούν ότι κάνω λάθος, αλλά από όσο γνωρίζω η εν λόγω εταιρεία έχει χρεοκοπήσει και δεν είναι σε θέση ε, να πληρώσει αποζημίωση. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υπομειστεί όλο το βάρος. Θα μπορούσε να δοθεί βοήθεια μορφή δανεισμού ή υπό άλλη μορφή. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να δίνει λάθος μήνυμα προς τις επιχειρήσεις γιατί θα τους δίνουμε την εντύπωση ότι κάποιος άλλος θα αναλάβει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη δική τους δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό σε διάφορα προγράμματα που βρίσκονται εν εξελίξη και για τα οποία έχουμε διάφορες αμφιβολίες για την υλοποίησή τους. Ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή εάν θεωρεί ότι από αυτό το ατύχημα και την καταστροφή στην Ουγγαρία αυτά τα οποία βιώσαμε καθιστά ακόμη πιο απαραίτητη την οδηγία για τα εδάφη. Δεν θα πρέπει να προχωρήσει η οδηγία για τα εδάφη στο Συμβούλιο και να φτάσει στην ολοκλήρωσή της. Πιστεύω ότι είναι επίγουσα πλέον η ανάγκη να έχουμε σαφείς διατάξεις για την αποφυγή της μόλυνσης των εδαφών και να έχουμε διαδικασίες για την απορρίπανση των εδαφών. Και δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο για να γίνει αυτό παρά η οδηγία για τα εδάφη που είναι πλέον επίγον ε, να προχωρήσει η κατάσταση στην Ουγγαρία θα ήταν διαφορετική αν υπήρχε η οδηγία για τα εδάφη. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα είχε βοηθήσει η οδηγία για τα εδάφη την Ουγγαρία να αντιμετωπίσει ή να προλάβει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κρήτον. Κυρία Μπλάνκο, θέλετε να απαντήσετε εν συντομία στις ερωτήσεις που σας θέσαμε εκ μέρους της Επιτροπής μας. Thank you very much, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με, την επικινδυνότητα της α, ε, ερυθράς που πραγματικά γιατί δεν χαρακτηρίστηκε σαν επικίνδυνο απόβλητο να σας πω ότι η οδηγία για την επεξεργασία και την διάθεση αυτής των επικινδύνων ουσιών εφαρμόζεται. Όμως η Ουγγαρία θεωρεί ότι δεν είναι εφαρμόσιμη αυτή η οδηγία. Άρα αυτό είναι ένα από τα θέματα το οποίο θα παρακολουθήσουμε και ήδη στη συνάντηση με την Ουγγαρία διαβιβάσαμε το, τις απόψεις μας στην Ουγγρική κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα την ταξινόμηση, ένα ένα προκαταρκτικό ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν υπάρχει υποχρέωση από τα κράτη-μέλη να ταξινομήσουν την ερυθρά ύλη σαν ε, μη, σαν ε, επικίνδυνο απόβλητο. Σύμφωνα με τον κατάλογο υπάρχουν δύο δυνατότητες ε, για την ταξινόμηση. Καταρχάς τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν με βάση την σύσταση του απόβλητου κατά πόσο το απόβλητο αυτό θα πρέπει να ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο ή όχι. Εάν υπάρχουν ε, επικίνδυνα συστατικά σε αυτή την ερυθρά ύλη που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, τότε η ερυθρά ύλη θα πρέπει να χαρακτηριστεί σαν επικίνδυνη. Επίσης, ο κατάλογος αποβλήτων ε, προ... Ε, προβλέπει ότι κάποιες τοξικές ουσίες, οι ουσίες που πειράζουν αν θέλετε τον οργανισμό θα πρέπει να χαρακτηριστούν ε, ε, επικίνδυνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που πήραμε από τις Ουγγρικές Αρχές ε, βλέπουμε ότι με την πρώτη ανάλυση που κάνουμε τα, τα συστατικά τα οποία αποτελούν την ερυθρά ύλη είναι επικίνδυνα. Όμως επειδή είναι ιδιαίτερα πτυτική, πτυτικά αν θέλετε τα συστατικά αυτά, δεν θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ότι η, η ανάλυση αυτή, η πρώτη αυτή ανάλυση θα είναι και οριστική. Πάντως η πρώτη μας ανάλυση είναι ότι πρόκειται για ε, επικίνδυνο απόβλητο. Λοιπόν, μέσα στα, ε, στις άδειες του 2000, στην του, του IPPC του 2006, όντως αυτό ισχύει, αλλά δεν το είχαν ταξινομήσει έτσι. Έχουμε αρκετές νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν και που εφαρμόζονται. Μπορεί να μην ε, εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά επί του παρόντος δεν θεωρούμε ότι μπορεί οποιαδήποτε task force να προσφέρει κάτι παραπάνω στην κατάσταση ή στην μελέτη και την ανάλυση της κατάστασης. Επίσης θα ήθελα να απαντήσω και στο ερώτημα για παρόμοια ε, sites στην Ευρώπη, παρόμοιες τοποθετήσεις ε, ε, στην Ευρώπη. Έχουμε νέα μονάδες παραγωγής βοξίτου που προ... παράγουν τεράστιες ποσότητες βοξίτη. Έχουμε εννέα εγκαταστάσεις αλουμίνας που επεξεργάζονται αυτό το βοξίτη, ο οποίος είτε εισάγεται είτε εξορίσεται. Από αυτά τα εννέα δηληστήρια, αν θέλετε, οι εγκαταστάσεις ε, επεξεργασίας, Έχουμε στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ρουμανία, στην Ισπανία και στην Ουγγαρία. Δεν είναι μόνο ή στην Ουγγαρία. Υπάρχουν ε, έγγραφα διαθέσιμα για την διαχείριση και την επεξεργασία του βοξίτη επιτόπου. Ε, βλέπουμε τι γίνεται με τα απόβλητα, τι γίνεται με, το, με τα ορυκτά κτλ. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά τα στοιχεία. Επίσης ζητήσατε να σχολιάσουμε λίγο το θέμα της παρακολούθησης. Εάν δείτε την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές που πέρυσι το καλοκαίρι ε, υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε και υιοθετήθηκε πρόσφατα, οι απαιτήσει ε, για την επίβλεψη και την εποπτεία έχουν ενταθεί για να είμαστε σίγουροι ότι η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται και για αυτού του είδους εγκαταστάσεις εφαρμόζεται η νομοθεσία, άρα μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους ε, επιβλέψεις, έτσι ώστε να μην ε, επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Νομίζω ότι απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Θα σας ανακοινοποιήσουμε βέβαια και τις, την τελική ανάλυση, τα αποτελέσματα μάλλον της τελικής ανάλυσης ε, που έχουμε κάνει για τα θέματα αυτά, γιατί επί του παρόντος, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη μας, έχουμε προχωρήσει μόνο σε μια πρώτη ανάλυση. Ευχαριστώ κυρία μου για αυτές τις διευκρινήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλουμε να, να καταλάβουμε πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία και αν εφαρμόζεται γιατί καταλήξαμε σε αυτή την τραγική κατάσταση. Περνάω επομένως στο επόμενο θέμα μας που είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Πία Μπουτσέλα η οποία θα μας παρουσιάσει γενικά την κατάσταση για τις συνθήκες κατά τις οποίες εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή και μετά θα ξεκινήσουμε με τις διάφορες ερωτήσεις ξεκινώντας με την κρίση στην Καμπανία. Στο σημείο 4 γιατί ακριβώς είναι η κυρία Μπουτσέλα η οποία θα πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ούτως ή άλλως ε, για το, το ερώτημα υπαριθμών 7 συζητήσαμε χτες για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Η κυρία Μπουτσέλα ή Μπουσελά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στην Επιτροπή να παρουσιάσει ε, την ε, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου για το Περιβάλλον. Καταρχήν θα σας ενημερώσω για πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ε, παραβάσεων και θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια και δράσεις τις οποίες υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει το ρόλο των εθνικών δικαστών στην επιβολή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή εφαρμόζει μια πολιτική μεγαλύτερης διαφάνειας στην διαχείριση των θεμάτων παραβάσεων. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή ανακοινώνονται στον τύπο από τη στιγμή της αιτιολογημένης γνωμοδότησης και στη συνέχεια. Από το καλοκαίρι στον τομέα του περιβάλλοντος Έχουμε εκδώσει πάνω από 30 ανακοινοθέντα τύπου. Το λέω αυτό για να σας δώσω μία διάσταση του έργου της Επιτροπής και των αποφάσεων που λαμβάνονται στον τομέα αυτό. Τις αποφάσεις αυτές μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα μας στο Ευρώπα, αλλά θεώρησα ότι θα ήταν χρήσιμο να σας ε, παρουσιάσω εγώ τις πιο σημαντικές αποφάσεις ανατομέα. Στον τομέα των αποβλήτων είχαμε αρκετές αποφάσεις. Τον Οκτώβριο η Επιτροπή αποφάσισε ε, ε, να πάει την Ιταλία στο δικαστήριο για δεύτερη φορά για τη μη εφαρμογή μιας απόφασης του 2004 σχετικά με τον καθαρισμό διαφόρων χωματερών κοντά στο Μιλάνο. Η Επιτροπή ζήτησε από το δικαστήριο να επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα, ημερήσιο πρόστιμο 25.400 ευρώ και ένα συνολικό ποσό πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Άλλο ένα ε, θέμα με βάση το άρθρο 260 ε, αφορά και την Ελλάδα για την ε, μη εκτέλεση μιας απόφασης του 2005 για παράνομες χωματερές και πάλι που ανέρχονται σε εκατοντάδες. Και στις δύο περιπτώσεις ε, είναι ανησυχητική η κατάσταση, γιατί οι αποφάσεις είναι αποφάσεις ε, που, είναι, που υπάρχουν εδώ και έξι χρόνια στην περίπτωση της Ιταλίας, πέντε χρόνια στην περίπτωση της Ελλάδας. Είχαμε άλλη μια υπόθεση του άρθρου 260 κατά της Μάλτας, για το παράνομο κυνήγι, άλλο ένα θέμα στον τομέα της προστασίας της φύσης. Και εδώ η, το νομικό πλαίσιο που θα επέτρεπε το κυνήγι 25.000 πτηνών ετησίως δεν θεωρείται συμβατό με το κριτήριο της αναλογικότητας που έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια απόφαση που εξέδωσε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Στον τομέα του ύδατος υπάρχουν πάλι διάφορες υποθέσεις κατά αρκετών κρατών μελών για την μη ε, έγκριση σχεδίων διαχείρισης ε, ποταμών. Δέκα αιτιολογημένες γνώμες έχουν ε, σταλεί μέχρι τώρα και Επίσης, με βάση το άρθρο 260, έχει σταλεί μια πρώτη προειδοποίηση στο Λουξεμβούργο για την μη συμμόρφωση με προηγούμενες αποφάσεις του δικαστηρίου και συγκεκριμένα για την μη κατάλληλη επεξεργασία αποβλήτων σε διάφορες αστικές περιοχές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τέσσερα κρατημένα, αντίον τέσσερα, τέσσερα κρατών μελών έχει ασκηθεί διαδικασία, γιατί δεν τηρούν την ομοθεσία για τις οριακές τιμές για το PM10 και υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλες υποθέσεις για το ίδιο θέμα που επίσης ε, προωθούμε στο δικαστήριο. Ε, επιστολέ προειδοποίησης έχουν σταλεί στην Ισπανία και στην Πορτογαλία γιατί δεν έχουν εκτελέσει δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά την έλλειψη σχεδίων έκτακτης ανάγκης για ορισμένες εγκαταστάσεις όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας σε Βέζο και το ερώτημα που τέθηκε νωρίτερα τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη σχεδίων εκτάκτου ανάγκης στον τομέα αυτό. Το δικαστήριο από το καλοκαίρι και μετά έχει εκδώσει και άλλες σημαντικές αποφάσεις. Σε μια συγκεκριμένη απόφαση καταδικάστηκε η Αυστρία λόγω ελήψεων στον προσδιορισμό προστατευμένων περιοχών σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά. Σε μια άλλη υπόθεση, το δικαστήριο έκρινε ότι η Σουηδία και η Σλοβενία δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους για ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές άδειες για ορισμένες υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σας τα είπα όλα αυτά για να σας παρουσιάσω την ένταση εργασιών της Επιτροπής καθώς και την ανάγκη να συνεχίσουμε να προωθούμε την εκτέλεση των αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφόσον είμαστε θεματοφύλακες των συνθήκων. Πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το όργανο που εφαρμόζει παντού την ευρωπαϊκή ε, ε, περιβαλλοντική ε, νομοθεσία. Σε μια ανακοίνωση του 2008 για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τονίσαμε την ανάγκη να εντείνουμε τις δράσεις εφαρμογής επικεντρωνόμενοι σε θέματα τα οποία μπορούν να προσθέσουν αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι αρχές στα 27 κράτη-μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνε για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και αν οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν εκπληρούν τα καθήκοντά τους, οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους. Γιατί πρέπει να εφαρμόζουν και το κοινοτικό δίκαιο. Οι περισσότερες ε, υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή περιβαλλοντικού δικαίου θα μπορούσαν ε, να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά ε, σε εθνικό επίπεδο, πιο αποτελεσματικά από ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, όλο και περισσότερο επαφιέμεθα στους εθνικούς δικαστές για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι εθνικοί δικαστές έχουν ευρείες δικαιοδοσίες έρευνας, μπορούν να λάβουν προσωρινά μέτρα και όπου είναι απαραίτητο μπορούν να απευθύνουν προδικαστικά ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Λουξεμβούργο. Επίσης, οι εθνικοί δικαστές ε, είναι νομικοί υψηλού κύρους ε, και έχουν και συνταγματικές εγγύησεις σε όλα τα κράτη-μέλη για το ρόλο που αναλαμβάνουν. Με βάση την προσέγγιση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθως ε, δεν ε, ε, συνεχίζει υποθέσεις παραβιάσεων όταν εκκρεμούν υποθέσεις σε εθνικά δικαστήρια. Πρόσφατα, το Σεπτέμβριο, είχαμε μια τέτοια περίπτωση όταν η ετήσια έκθεση, η 27η έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή. Στην έκθεση μας αυτή, αναφέρεται ότι η Επιτροπή δεν θα αναλαμβάνει παράλληλη δράση όταν η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει τη δημιουργία εθνικών μηχανισμών για δικαστική επανεξέταση. Αυτός ο μηχανισμός απαιτείται σύμφωνα με κάποιες υφιστάμενες οδηγίες, όπως είναι η οδηγία για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη η οδηγία για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η οδηγία για τις ε, βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Βασιζόμαστε όλο και περισσότερο σε εθνικές ε, δικαστικές διαδικασίες για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου και αυτό έχει γίνει με την ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και Εθνικών Δικαστών. Υποστηρίζουμε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Δικαστών για το Περιβάλλον στις προσπάθειες που καταβάλει να προωθήσει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τότε που, άρχισε, από τότε που δημιουργήθηκε το 2004. Επίσης, συνεργασία με δικαστές έχουμε και με σύνδεση Ευρωπαίων ε, Διοικητικών Δικαστών και εθνικών δικαστηρίων. Υπάρχουν ε, και προγράμματα κατάρτισης με διάφορα ε, σεμινάρια τα οποία αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση για το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο στους κέριους τομείς, ιδίως για την προστασία της φύσης και για τα απόβλητα και προσπαθούμε να βοηθούμε τους εθνικούς δικαστές για να εφαρμόζουν αυτήν την νομοθεσία στην πράξη. Αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει ένα φόρουμ για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων μεταξύ εθνικών δικαστών. Οργανώσαμε και μία διάσκεψη για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου με δικαστές και εισαγγελείς από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η διάσκεψη αυτή είχε πάνω από 150 συμμετέχοντες, δικαστές και εισαγγελείς από Ισπανία και Πορτογαλία, έλαβε χώρα στη Σεβίλη πριν από λίγες μέρες. Άλλη μια παρόμοια διάσκεψη θα οργανωθεί στην Ιταλία του χρόνου. Ιταλοί και Ρουμάνοι δικαστές και εισαγγελείς θα συμμετάσχουν στην διάσκεψη εκείνη. Παράλληλα, Προσέχουμε ιδιαίτερα την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Όρχους για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Η πρόταση της οδηγίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα παραμένει σε επίπεδο συμβουλίου σε αδιέξοδο και αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Όμως κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας περιλαμβάνουν διατάξεις για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως ανέφερα προηγουμένως, τη οδηγία για την, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οδηγία για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αποτελεσματικά και αυτό για μας αποτελεί προτεραιότητα. Εις επίμετρον. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν τους εθνικούς δικαστές να εκπληρώσουν πιο αποτελεσματικά το ρόλο τους για το περιβάλλον. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα σύστημα πολλαπλών επιπέδων για τη διακυβέρνηση και ο δικαστικός μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί σωστά σε εθνικό επίπεδο και αυτό είναι αποτελεσματική προϋπόθεση για να διασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής μας νομοθεσίας και του περιβάλλοντος συνολικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας αυτή τη τόσο πλήρη. Θα δούμε πρώτα τις ερωτήσεις 4 με 12 που έχουν να κάνουν με τα απόβλητα, με την κρίση αποβλήτων στην καμπανία. Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα παρέμβουν οι άλλοι συνάδελφοι. Συνδυάστε αυτά τα δύο σημεία 4 και 12 παρακαλώ. Ναι. Στις 4 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επεφάνθηκε ότι η Ιταλία παραβίασε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν δημιούργησε στην καμπανία δίκτυο εγκαταστάσεων το οποίο να είναι επαρκές ώστε να διασφαλίζει τη διάθεση των αστικών αποβλήτων κατά τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αυτή είναι η, αυτό είναι η απόφαση. Παρ' όλα αυτά η Ιταλία δεν έχει έκτοτε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Στις 23 Οκτωβρίου που μας πέρασε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ κοντά στην κρίση που είχαμε το 2007 και η οποία μας ε, οδήγησε στο να ξεκινήσουμε διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας. Τα επικίνδυνα απόβλητα αναμειγνύονται και διατίθενται μαζί με οικιακά ή και οργανικά απόβλητα κατά παράβαση της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα και της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό που έχω να πω για αυτήν την ε, γενική ερώτηση είναι το εξή. Ότι ελέγχουμε προσεκτικά το τι κάνουν οι Ιταλικές αρχές για να ανταποκριθούν στην απόφαση. Υπήρξαν πολλές ε, συναντήσεις που είχαμε με τις περιφερειακές αρχές και έχουμε ήδη στείλει δύο επιστολές στην Ιταλία προκειμένου να δούμε τι κάνουν μετά από την απόφαση του δικαστηρίου. 21 και 22 Νοεμβρίου πιο συγκεκριμένα πήγαμε στην Καμπανία. Κατά την επίσκεψή μας αυτή συναντηθήκαμε με περιφερειακές αρχές εκεί. Όπως επίσης Συναντήσαμε και περιβαλλοντικούς συμβούλους από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Φύγαμε μόνο σε μία μονάδα καύσης ε, εκεί. Στο Τερζίνιο και είδαμε πώς διοχετεύονται 8.000 τόνοι αποβλήτων. Η αποστολή μας πάντως επιβεβαίωσε, και ακριβώς αυτό είπαμε και στον Επίτροπό μας, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να συμμορφωθεί η περιοχή με την απόφαση του δικαστηρίου δεν υπάρχουν ακόμα. Παρόλο που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της απόφασης. Πρώτα απ' όλα, η καμπανία πρέπει να υιοθετήσει κατεπηγόντως ένα νέο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Εμείς θεωρούμε ότι προκειμένου να αποφύγουμε επαναλαμβανόμενες κρίσεις, αν και αυτήν που είχαμε το 2007, η τεράστια κρίση επίσης που ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε ή και άλλες όπως εκείνη με τα σκουπίδια που εξακολουθούμε να βλέπουμε στους δρόμους της Νάπολης, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα διαρθρωτικό σύστημα διαχείρισης, συλλογής, ε, απορριμμάτων και διαχωρισμού απορριμμάτων επίσης. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο να συμμορφώνεται απόλυτα στις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής ε, Νομοθεσίας για το Περιβάλλον. Προτεραιότητα βέβαια πρέπει να δοθεί στην ιεράρχηση των αποβλήτων 12 Δεκεμβρίου θα είμαστε έτοιμοι με τη νέα οδηγία. Θα αρχίσει να ισχύει η νέα αυτή η οδηγία πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην μείωση των αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίησή τους και στην ανακύκλωσή τους. Δεύτερον, το νέο σχέδιο διαχείρισης πρέπει να διασφαλίσει και εφαρμογή χωριστής συλλογής σε ολόκληρη την περιοχή, κυρίως στην πόλη και στην περιοχή της Νάπολης που δεν υπάρχει ακόμα πλήρως. Γιατί εκεί έχουμε πάνω από 50% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής της Καμπανίας. Το σχέδιο διαχείριση πρέπει να προσφέρει ε, καλές δυνατότητες κομποστοποίησης των αποβλήτων. Πρέπει να είναι έτοιμο σύντομα, μια που μιλάμε για 8 εκατομμύρια τόνους. Α, συγγνώμη, 8 εκατομμύρια που πάνε σε διάφορα σημεία στην καμπανία. Έχουμε λοιπόν υπογραμμίσει τα στοιχεία αυτά και όταν πήγαμε στην καμπανία την προηγούμενη εβδομάδα. Οι περιφερειακές αρχές μας υποσχέθηκαν ότι θα υποβάλουν στην Επιτροπή σχέδιο για το νέο πρόγραμμά τους και ότι θα υιοθετήσουν σε περιφερειακό επίπεδο, στην περιφερειακή κυβέρνηση, το σχέδιό τους μέχρι τον Απρίλιο που μας έρχεται. Εμείς υπογραμμίσαμε ότι το σχέδιο αυτοδιαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας διάφανης διαδικασίας στην οποία να συμμετέχουν όλοι προκειμένου το σχέδιο αυτό να έχει περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, πρώτα απ' όλα η κρίση αποβλήτων θα επανέλθει ξανά και ξανά. Είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό. Έπειτα θα υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και κίνδυνος για καταστροφές στο περιβάλλον. Το δικαστήριο Ίσως σε αυτή την περίπτωση, ε, μάλλον έχει αναφερθεί σε αυτό με την απόφαση του το δικαστήριο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον δεν υπάρχει σχέδιο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πάει και πάλι στο δικαστήριο. Με αποτέλεσμα επιβολής προστίμου για την καμπανία. Συνεπώς, θα αξιολογήσουμε το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που θα μας στείλει πριν από τα τέλη της χρονιάς η περιοχή. Και στη συνέχεια θα ελέγξουμε την κατάσταση προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο αυτό. Η απόφαση τώρα για το πώς και πότε να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία του άρθρου 260 για αυτή την περίπτωση θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο, από το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και από την ίδια την εφαρμογή, κατά πόσο θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Όσον αφορά τώρα το θέμα, κατά πόσο τα απόβλητα αυτά ανακατεύονται με οικιακά απόβλητα, εμείς δεν έχουμε αποδείξεις. Τον έλεγχο για αυτό το θέμα τον έχει το κράτος. Είναι εθνική αρμοδιότητα. Όσον αφορά τώρα το ότι η χωματερή είναι παράνομη, επειδή είναι σε ένα εθνικό πάρκο, το γεγονός αυτό από μόνο του δεν παραβιάζει την οδηγία για τους χώρους υγειονομικής ταφής, γιατί δεν αναφέρεται τέτοια διάταξη στην ίδια την οδηγία. Όσον αφορά τώρα τη υπόνοιες ότι το Τερτσίνιο είναι χώρος που παραβιάζει την οδηγία, είναι κάτι το στην διαδικασία επιπαραβάση που έχει ανοίξει κατά της καμπανίας. Εμείς γνωρίζουμε ότι στην Καμπανία υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των αποβλήτων. Είμαστε πεπισμένοι ότι όλα αυτά τα προβλήματα αποτελούν τη συνέπεια έλλειψης ενός κανονικού, ενός καλού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που θα έπρεπε να υπήρχε. Και γι' αυτό και επικεντρωθήκαμε στις διαδικασίες μας ήδη από την αρχή στην διαχείριση των οικιακών αποβλήτων. Και γι' αυτό επίσης με την απόφασή του το δικαστήριο επέμεινε για το ότι η Ιταλία πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει όσο γίνεται πιο γρήγορα ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Νομίζω ότι έτσι σας έδωσα μια συνολική εικόνα της κατάστασης πραγμάτων όπως έχει σήμερα στην καμπανία. Αν έχετε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν να συνεχίσουμε αγαπητοί συναδελφοί να σας πω ότι στην αίθουσά μας βρίσκεται η Ιταλική τηλεόραση. TG24 είναι μια ιδιωτική, ένα ιδιωτικό κανάλι τηλεόρασης. Ε, δεν ξέρω αν έχετε καμία αντίρρηση ε, το κανάλι αυτό να μαγνητοσκοπήσει τις, ε, τις συζητήσεις μας. Λοιπόν, θα ήθελα να χαιρετήσω και την, ε, παρουσίαση, την παρουσία της κυρίας Μαντζόνη, που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών και δίνω το λόγο στην κυρία Τζιλ Evans, που είναι η πρώτη στον κατάλογο μου και μετά θα συνεχίσουμε. Jill Evans. Δεν θέλει. Η Ζητήτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπουτσέλα για τις διευκρινήσεις που μας έδωσε. Τον Μάιο, τον Απρίλιο-Μάιο του 2010, είχαμε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών ε, στην Καμπανία για να απαντήσουμε σε κάποιες, αναφορές, που είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή μας για τους ε, κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία. Επισκεφθήκαμε τις χωματερές, ε, τον αποτεφρωτή, είδαμε τα απόβλητα, είδαμε τις παράνομες χωματερές το πρόβλημα είναι ότι αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι υπήρχαν πολλά σχέδια στο παρελθόν και καλά σχέδια. Και το πρόβλημα στην καμπανία είναι η εφαρμογή. Και το είπατε και εσείς πολλές φορές ε, ότι το θέμα είναι η εφαρμογή. Εσείς ελέγχετε την κατάσταση, παρακολουθείτε την κατάσταση, μιλήσατε για τη διαδικασία του άρθρου 260 και είπατε για το ότι κατά πόσον θα ενεργοποιήσετε τη διαδικασία του άρθρου 260 εξαρτάται από το περιεχόμενο του σχεδίου, από την ποιότητα του σχεδίου, από, την, ε, από το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το σχέδιο και από την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος. Αυτό το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι. Μιλάμε για το χρονοδιάγραμμα της δικαστικής απόφασης Μαρτίου. Μιλάμε για το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το σχέδιο της καμπανίας ή μιλάμε για το δικό σας χρονοδιάγραμμα. Αν λέτε ότι η εφαρμογή ε, και ο έλεγχος ας πούμε των επικινδύνων επιβλήτων, των οικιακών αποβλήτων. Είπατε ότι ο έλεγχος ανήκει σε εθνικό επίπεδο αλλά χρειαζόμαστε στοιχεία ε, που προέρχονται από τον έλεγχο για να δούμε κατά πόσο η οδηγία εφαρμόζεται σωστά. Επομένως, πώς θέλ προβλέπετε να τα συντονίσετε όλα αυτά. Πώς μπορείτε να δείτε ότι η οδηγία εφαρμόζεται σωστά εάν ο έλεγχος ε, για την εφαρμογή της βρίσκεται σε εθνικά χέρια. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Είπατε ότι Είπατε επίση ότι για το Τερτσίνιο ότι η παρουσία χωματερή σε ένα εθνικό πάρκο δεν προβλέπεται καν στην οδηγία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κενό τη οδηγία. και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και θα το κάνω εγώ στο Κοινοβούλιο για να καλύψουμε το κενό αυτό. Επίσης, ο Επίτροπος Ποτότσνικ κάνει μια επίσκεψη στην περιοχή, άκουσα, Άκουσα ότι θα δει την κατάσταση ο ίδιος με τα μάτια του το Φεβρουάριο. Θα επισκεφθεί τη χωματερή όντως. Ε, θα γίνει κάτι για να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία, τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλικής είναι η κυρία Μαντσόνη από την Επιτροπή Αναφορών. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ γιατί μια, έστω και αν δεν αποτελώ μέλος της Επιτροπής μου δίνεται το λόγο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ερώτημα που μας απασχολεί σήμερα και απασχολεί την Επιτροπή σας δεν αφορά μόνο την χώρα μου, αλλά και γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, με το οποίο ασχοληθήκαμε στην Επιτροπή Αναφορών. Το είπε και η συνάδελφος Μέρκες. Θέλω να πω, καταρχάς, ότι ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή, γιατί, την Κομισιόν δηλαδή, ε, διότι παρακολουθεί το πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μαστίζει εδώ και χρόνια την καμπανία και ανησυχεί αρκετά την ε, Ιταλία. Είναι ένα παλιό θέμα, ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί και επιδεινώνεται με την πάροδο του έτους, τον, ε, με την των ετών. Η κυρία Βουτσέλα είπε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που έγινε πριν από λίγες μέρες ε, στην Καμπανία και στην περιοχή της Νάπολης κυρίως, ε, είδε με τα μάτια της ότι όντως ε, ε, υπάρχει λόγος ανησυχίας, ότι υπάρχουν ακόμα τα σκουπίδια στους δρόμους και ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Για μας ε, είναι σκόπιμο να υπάρχει το προσεκτικό μάτι της Ευρώπης πάνω από την Ιταλία διότι όλα τα, όλες οι υπηρεσίες που, που αφορούν την διαχείριση των αποβλήτων στην Ιταλία λειτουργούν, πρέπει να λειτουργούν έγκαιρα. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι σε όλες τις ακροάσεις που αφιερώσαμε στο θέμα. Ακούσαμε και, του, και υπευθύνους από την καμπανία και άκουσα επίσης ε, και την συζήτηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της περιοχής ε, με τους ε, επιτρόπους και ακούσαμε ότι έχουν αναλυφθεί σημαντικές δεσμεύσεις όχι μόνο ε, αυτά που είπε η καθηγήτρια κυρία Μπουτσέλα για το χρονοδιάγραμμα, ότι θα έπρεπε το σχέδιο να υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το προσωρινό και το οριστικό το επόμενο τρίμηνο, αλλά ε, μιλάγαμε, έχουμε ακούσει και για δεσμεύσεις που θα πρέπει να, αναλάβει η, να αναλάβουν οι τοπικές αρχές και που αφορούν το περιβάλλον. Παραδείγματο χάρη ε, ένα σχέδιο για, την, για τον διαχωρισμό, συλλογή και διαχωρισμό των αποβλήτων, ε, η επαναχρησιμοποίησή τους Αυτά είναι θέματα που ελπίζω ότι θα παραμείνουν στο σχέδιο. Επομένως, εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή όχι μόνο ο σεβασμός των ημερομηνιών, αλλά και ο σεβασμός του περιεχομένου του σχεδίου, έτσι όπως ε, ε, έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Αναφορών. Επίσης, και η κυρία Μέρκης, η οποία ήταν υπεύθυνη και επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, της Επιτροπής Αναφορών στην Καμπανία, θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Γιατί η κυρία Μπουτσέλα μιλήσε για τις ε, προθεσμίες, ε, τις προθεσμίες που έχουν αποφασιστεί αλλά εδώ μιλάμε για προθεσμίες 12 και 24 μήνες για την εφαρμογή της ε, απόφασης ε, του δικαστηρίου, δηλαδή 12 και 24 μήνες για να υιοθετηθεί το σχέδιο ε, το οποίο προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή το δικαστήριο καταδικάζει την Ιταλία όχι μόνο διότι δεν εφάρμοσε εγκαίρως το σχέδιο, αλλά γιατί δεν το εφάρμοσε εγκαίρως το σχέδιο το οποίο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το περιεχόμενο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Εδώ θα ήθελα να καθέσω και ένα ερώτημα, το οποίο δεν το κάνω όμως, διότι το είπε και η κυρία Μέρκης ε, για την ε, διαδικασία που θα ξεκινήσει με βάση το άρθρο 260. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη στην Ιταλία με, ε, με τον τύπο φαινόταν ότι η χώρα μας και πιο συγκεκριμένα η καμπανία αποτελούσε αντικείμενο νέας διαδικασίας επί παραβάση ενώπιον του δικαστηρίου. Η καθηγήτρια κυρία Μπουτσέλα ε, απήντησε ήδη και θα το διευκρινίσει ακόμα περισσότερο ότι η διαδικασία του άρθρου 260 μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο και εφόσον αυτό το σχέδιο το οποίο έχουν, ε, έχουν ε, προαναγγείλει οι τοπικές αρχές της Καμπανίας δεν υιοθετηθεί μέχρι τον Μάρτιο και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε ξανά στο δικαστήριο. Τώρα, επίσης ε, καταλαβαίνω την έκπληξη της ε, συναδέλφου κυρίας Μέρκης ε, όσον αφορά το ότι δεν είναι αντιφατικά, αντιφατικό να υπάρχει μια χωματερή σε ένα εθνικό πάρκο, σε ένα πάρκο, εθνικό πάρκο και ότι η ύπαρξη μιας χωματερής σε εθνικό πάρκο δεν παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Εμεί θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν προφανή παραβίαση τη ε, κοινωτική νομοθεσία, αλλά φαίνεται, μα είπε η κυρία Μπουτσέλο, ότι δεν υπάρχει ε, τέτοια πρόβλεψη στην ε, κοινωτική νομοθεσία. Τώρα βέβαια από τη μία πλευρά ε, είναι θετικό το στοιχείο διότι αυτό σημαίνει ότι η Ιταλία δεν έχει παραβιάσει την κοινοτική νομοθεσία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά από την άλλη πλευρά θα ζητούσα και εγώ ε, από την ε, Κομισιό να παρακολουθήσει με περισσότερη προσοχή τέτοιου είδου περιπτώσεις διότι εδώ μιλάμε και για προστασία του περιβάλλοντο και ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε και τις ζώνες ε, που είναι ήδη προστατευμένες. Όταν μιλάμε το εθνικό πάρκο, για το Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου, ε, είναι περίεργο από τη μία πλευρά να το προστατεύουμε το Εθνικό Πάρκο και από την άλλη πλευρά να μην αποκλείουμε την εγκατάσταση χωματερών. Και ολοκληρώνω την παρέμβασή μου εκφράζοντας την διαθεσιμότητά μου να συνεργαστώ με την Επιτροπή για να επιταχύνουμε τους χρόνους και τις προθεσμίες ε, επικοινωνίας ε, ανάμεσα στις ε, τοπικές αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να διευκολύνω όσο δυνατόν περισσότερο των ε, τοπικών αρχών για να μπορέσουν να σεβαστούν τις προθεσμίες που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ένα από τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τριβελίν είναι ο επόμενος ομιλητής, μετά ο κύριος Πρόδη, Αρσένης και Ρώση. Ε, σας παρακαλώ μόνο να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε και άλλα σημεία και μέχρι το μεσημέρι πρέπει να βιαστούμε λίγο. Κύριος Ριβελίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπουτσέλ. Εγώ δεν παίρνω το λόγο μόνο σαν Ιταλός βουλευτής, αλλά σαν, ε, σαν αυτή ε, ε, γιος αυτής της μαρτυρικής γης που κάποτε ήταν κομμάτι και είναι ακόμα δηλαδή της Μεγάλης Ελλάδας και που απασχολεί την Ευρώπη για ένα τόσο δραματικό θέμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο όταν μιλάει για ένα χρονοδιάγραμμα, για το ότι θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να υποβληθεί ένα προκαταρκτικό σχέδιο, ότι θα πρέπει να, σεβαστεί, να σεβαστούν τοπικές αρχές ε, της καμπανίας, τα, τις διατάξεις του σχεδίου αυτού, ε, συμφωνώ με τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν, διότι είναι παράλογο το 2010 να υπάρχει μια κατάσταση τόσο τραγική. Κατανοώ απόλυτα ποιο είναι το καθήκον της ε, Επιτροπής, κατανοώ απόλυτα ότι αναλύονται όλες αυτά τα στοιχεία ε, και κατανοώ απόλυτα ότι οι δικαστές πρέπει να τιμωρήσουν ε, τις ε, ανίκανες τοπικές αρχές. Μετά πρέπει να δούμε βέβαια και ποιος είναι ουσιαστικά υπεύθυνος, ποιο, έχουν, ποιοι έχουν αποφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν είναι το θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι λείπει από την έκθεση της Επιτροπής κυρίας Μπουτσέλη είναι πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Εάν είμαστε εδώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να μην βοηθήσουμε μία κοινότητα η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ε, δεν μπορούμε μόνο γραφειοκρατικά να εκτιμούμε την κατάσταση. Δεν μπορούμε απλώς και μόνο να προβλέπουμε ε, κυρώσεις εναντίον της Ιταλίας και της Καμπανίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια για πάντα τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε αυτή την κρίση. Διότι η Καμπανία αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και άκουσα και, την, τον πρόεδρο της Επιτροπής, της, συγγνώμη, και τον πρόεδρο της ε, περιφέρειας, της περιοχής, που είναι και αυτός ιδιαίτερα ανήσυχο και ε, ε, πρέπει να σεβαστεί και τις, τις προθεσμίες που μας παρουσίασε η κυρία Μπουτσέλα. Και εγώ ρωτώ, υπάρχει ένα πρόγραμμα για τους Ευρωπαίους πολίτες στην Καμπανία. Στην Επιτροπή Αναφορών εγώ φωνάζω, φώναξα σαν πολίτης ε, αυτής της περιοχής ε, διότι εδώ είμαστε και κερατάδες και δαρμένοι, διότι το λένε και στην καμπάνια αυτό από ό,τι φαίνεται. Και όχι μονάχα στην Ελλάδα. Ε, διότι τα χρήματα τα οποία δίνονται για, την, για όλα αυτά, τα εισπράττει κάποιος που πάνε όμως δεν ξέρουμε. Και αντί να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τα λεφτά, τιμωρούμε τους πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες της καμπανίας. Επομένως, ζητώ από την κυρία Μπουτσέλα, υπάρχει θέληση από πλευρά της Κομισιόν να δει τα θέματα με έναν άλλον τρόπο και όχι μονάχα ε, από, την, ε, από τη σκοπιά της επιβολής κυρώσεων και ποινών και μία συγκεκριμένη ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Στην πρώτη παρέμβαση της κυρίας Μπουτσέλλα ε, ακούστηκε ότι η Ιταλία θα τιμωρηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κάποιες χωματερέσεις στο Μιλάνο. 22.000 ε, ευρώ την ημέρα. Μη δώσει και κάποιες ενδείξεις για το, θέμα, για το θέμα αυτό. Γιατί και εκεί θέλω να ξέρω. Υπάρχει μια Ιταλική αλληλεγγύη και μια ευρωπαϊκή ελληνική παράλληλα. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κ. Βιτόριο Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι επεπισμένος, όπως και οι συνάδελφοί μου, ότι είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς τόσο κακά πράγματα για την Ιταλία. Αλλά δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω το δαχτυλό μα. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ε, κατάματα. Επομένως, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ιταλία όπου ε, τα αντίστοιχα πράγματα γίνονται με τον σωστό τρόπο. Όταν ήμουνα πρόεδρος της ε, περιοχής ε, της περιφέρειας της Μπολόνια, υλοποιήθηκαν ε, σημαντικά έργα υποδομής στο επίπεδο συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων. Είχαμε έναν μεγάλο αποτεφρωτή και τρεις χωματερές υποστήριξης, αν θέλετε. Άρα υπάρχουν τρεις χιτά. Υπάρχουν ε, οι δυνατότητε στην Ιταλία, υπάρχουν οι υποδομές στην Ιταλία και θα πρέπει να αναλάβουμε μία δέσμευση εδώ για να υπάρξει αυτή η αλληλεγγύη που λείπει και από την Ιταλία την ίδια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει να ε, καθησυχάσουμε, να επιβεβαιώσουμε τους υπευθύνους ότι υπάρχουν οι πόροι. Διότι οι συνάδελφοι, φίλοι, είναι δύσκολο να δεχτούν ότι υφίσταται μια τέτοια κατάσταση. Όμως πιστεύω ότι η χώρα θα βρει τους απαραίτητους πόρους για να, και να βρει μια κατάλληλη λύση. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ύπαρξη του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ασένης. Thank you very much, I would like to ask the Commission whether this... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε και μια απάντηση για το Natura 2000 δίκτυο. Δεν ξέρω αν θα απαντήσετε σε αυτό πριν συνεχίσουμε με άλλες ερωτήσεις. Για το θέμα αυτό, οι πληροφορίες μου είναι ότι τμήμα του Ιταλικού Εθνικού Δρυμού στο Βεζούβιο είναι τμήμα του Natura 2000 του δικτύου. Τώρα, η ε, ε, ε, υπάρχουσα χωματερή στο Τερτσίνιο, στο άκρο του Εθνικού Δρυμού, δεν γνωρίζω αν είναι τμήμα της περιοχής Natura 2000. Νομίζω πως δεν είναι όμως. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω από την απάντησή σας ότι τέτοιες χωματερές επιτρέπεται να υπάρχουν σε περιοχές Natura 2000. Αν όντως επιτρέπεται, νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα. Και θα έπρεπε να εξετάσουμε τι επικίνδυνες δράσεις διεξάγονται, που είναι επικίνδυνες και για τη βιοπικιλότητα και τι πρέπει να αλλάξει. Αν όντως λοιπόν επιτρέπετε, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους άλλους συναδέλφους που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον ε, κύριο Αρσένη. Ο κύριος Ορέστε Ρώση είναι ο επόμενος ομιλητής. το θέμα των αποβλήτων της ε, καμπάνιας ε, και των ε, κατοίκων της Νάπολης δεν είναι ένα καινούριο θέμα. Εδώ και δεκαετίες λόγω, δεκαετίες λόγω κακής διαχείρισης δεν κατάφερναν να, να απορροφήσουν τα απόβλητά τους και πριν από δύο χρόνια ε, ε, και, στη Λομβαρδία και στο Πιεμόντε άνοιξαν νέες χωματερές για να απορροφήσουν τα, απόβλητα τα πόβλητα της ε, καμπανίας. Όμως, να, να, διευκρινίσω ότι οι κερατάδες και δαρμένοι δεν είναι οι πολίτες της Καμπανίας, είναι οι πολίτες της υπόλοιπης Ιταλίας που αναγκάζονται να πάρουν τα απόβλητα τα δικά τους. Λοιπόν, υπάρχουν, θα πρέπει να παρέμβει το κράτος και όταν υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος αγαπητέ Κρήτονα και άλλοι συνάδελφοι λοιπόν, εάν υπάρχουν προβλήματα με, τις, τα απόβλητα τα παίρνουν από εκείνη την περιοχή και τα πηγαίνουν σε κάποιο άλλο σημείο όντως το Τερτσίνιο είναι κοντά στο Εθνικό Πάρκο όπως είναι κοντά και μπορούν να το βάλουν να, να πάνε εκεί τα απόβλητα γιατί είναι κοντά και πρέπει να μπορούσαν να πάνε γρήγορα Άρα θα πρέπει ούτως ή άλλως οι τοπικές κυβερνήσεις, θα πρέπει και γενικότερα οι κυβερνήσεις, θα πρέπει οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να φτιάχνουν και χωματερές και αποτεφρωτές κτλ. Διότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει η Κομισιόν να, επιβληθεί, να επιβάλλει κυρώσεις. Αλλά τις κυρώσεις αυτές θα πρέπει να τις πληρώσουν οι τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνε και όχι οι εθνικές κυβερνήσεις και να μην πληρώνουμε εμείς που ε, πήραμε τα, τα απόβλητα εδώ 20 χρόνια αυτέ οι τοπικέ αρχέ τη Καμπανία που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα δικά του απόβλητα τα μοιράζουν σε όλη την υπόλοιπη Ιταλία. Και μετά όλη η υπόλοιπη Ιταλία πληρώνει. Αγαπητέ, αγαπητοί ε, εκπρόσωποι τη Κομισιόν, μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν είμαστε και πολύ ε, ικανοποιημένοι από αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό καλώ ε, την Κομισιόν να καταβάλει κάθε την προσπάθεια έτσι ώστε το σχέδιο αυτό να εκπονηθεί, να ασκήσετε πίεση στις τοπικές αρχές ότι θα πρέπει να εφαρμόσει το, το σχέδιο αυτό, διότι εάν τυχόν δεν το εφαρμόσει, αυτές οι κυρώσεις θα επιβληθούν. Και τις κυρώσεις αυτές θα πρέπει να πληρώσουν οι τοπικές αρχές που δεν θα να κάνουν τη δουλειά τους. E, e- Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρώση. Ο κύριος Τσουμπάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, να εξετάζουμε το θέμα κάπως αντικειμενικά. Είναι μια κατάσταση που κρατάει, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι πολίτες των οποίων το δικαίωμα στην υγεία πρέπει να διαφυλέξουμε. Το δικαίωμα στην υγεία νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε μια χωματερή η οποία βρίσκεται σε μια ζώνη που έχει κάποιους περιβαλλοντικούς ε, περιορισμούς. Και η Κομισιό και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο γενικότερα λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ταυτόχρονα όμως πέραν αυτού του αντικειμενικού στοιχείου υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος ε, Ρώση στην διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι για χρόνια ολόκληρα από την Βόρεια Ιταλία και από την Βόρεια Ευρώπη ερχόντουσαν φορτηγά τοξικών αποβλήτων τα οποία ακόμα βρίσκονται θαμμένα σε κάποιες ε, ε χωματερές παράνομες τις οποίες διαχειρίζεται παράνομα η καμόρα και η μαφία. Είναι ένα θέμα του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, να ξεκινήσουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες τις οποίες εξήγηλε η Κομισιόν σήμερα. Εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει, διότι είδαμε ότι υπάρχουν ε, και υποσχέσεις ε, του Πρωθυπουργού Μπερλουσκόνη, ο οποίος είπε θα τα, θα τα λύσω όλα τα, την προηγούμενη εβδομάδα είπε θα το λύσω σε 15 μέρες. Την προηγούμενη εβδομάδα είπε σε 3 μέρες θα το λύσω το πρόβλημα. Λοιπόν, Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να, σεβόμαστε ένα τέτοιον άνθρωπο ο οποίος ε, ε, δεν ξέρω πώς λειτουργεί τέλος πάντων. Κάποιος πρέπει να αναλάβει τα ενία, κάποιος πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει και να επιβάλλει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην καλύτερη θέση. E, Ευχαριστούμε. Επόμενος ή μάλλον πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή, ο κύριος Ριβελίνη ζήτησε το να μιλήσει. Μόνο μισό λεπτό, Πρόεδρε, για να υπενθυμίσω ότι η τοπική κυβέρνηση της Καμπανίας εξελέγει πριν από έξι μήνες και πρέπει να ξέρουμε ποιος φέρει τις ευθύνες. Ναι, αυτό είναι σωστό. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να βοηθήσουμε και αυτή τη νέα τοπική κυβέρνηση που νομίζω ότι έχει έρθει σε επαφή με την Κομισιόν και την κυρία Μπουτσέλα. Και να απαντήσω στον φίλο κύριο Ρώση, φίλο και συνάδελφο Ρώση, να υπενθυμίσω ότι αν οι τοπικές αρχές πρέπει να πληρώσουν για τις δικές τους ζημιές, ε, Ας πληρώσουμε και αυτά τα, αυτές τις κυρώσεις ε, που μας ε, θύμισε η κυρία Μπουτσέλα για τις χωματερές στο, στο Μιλάνο και στη Λομβαρδία και ε, ας πληρώσουν και όλες αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις της, του Βορρά που χρησιμοποίησαν την καμπάνια σαν χωματερή τους. Λοιπόν, ας το δούμε και αυτό. Είμαστε 20, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν 27 κοινότητες. Δεν, εάν θέλουμε να λειτουργήσουμε ενιαία, δεν πρέπει να, ε, δεν πρέπει να λειτουργούμε ως αν να υπάρχουν πολίτες ε, διαφόρων κατηγοριών, πολίτες Α, Β και Γ, διότι αλλιώς δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Ριβελίνη. Τώρα. Κύριε Μπουτσέλη. Mm. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια και η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έγιναν στα Ιταλικά. Θα απαντήσω και εγώ στα Ιταλικά και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Αρσένη που είμαι σίγουρη θα καταλάβει τι θα πω. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να διευκρινίσω ότι οι απαντήσεις μου αφορούσαν μόνο αυτό το οποίο, αυτά τα οποία ελέγχθησαν, ε, αυτά τα οποία και αυτά τα οποία είναι αρμοδιότητες της Κομισιόν. Υπάρχουν άλλα θέματα για τα οποία δεν είναι αρμόδια η Κομισιόν, άρα δεν μπορώ να τα σχολιάσω εγώ. Τώρα θα ήθελα να απαντήσω καταρφάς στην κυρία Μέρκης, η οποία ε, λείπει, αλλά θα της διαβιβάσουν ελπίζω την απάντηση. Ρώτησε συγκεκριμένα είπε για να αξιολογήσουμε την διαδικασία του άρθρου 260 η Κομισιόν θα στηριχθεί στο περιεχόμενο στα χρονοδιαγράμματα και στην ε, εφαρμογή και στο σεβασμό του προγράμματος διαχείρισης των αποβλημάτων. Και ήθελε να ε, ξέρει τι εννοούσα όταν είπα για χρονοδιαγράμματα, για προθεσμίες και νομίζω ότι και η απάντηση αυτή θα ισχύσει και για τις άλλες ερωτήσεις που ακούστηκαν. Καταρχάς, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι μια απόφαση, μια δικαστική απόφαση πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η εκτέλεση στη συγκεκριμένη περίπτωση της απόφασης του δικαστηρίου ε, αφορά τρία στοιχεία την υιοθέτηση του σχεδίου καταρχάς. Ε, το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, την εκτέλεση του σχεδίου και τρίτον την ε, διαχείριση, αν θέλετε, και την, ε, τον τρόπο που θα επεξεργαστούν αυτά τα σκουπίδια, αυτά τα απόβλητα. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε την ε, διάθεση αυτών των ε, συσκευασμένων σκουπιδιών, αν θέλετε, των 8 εκατομμυρίων τόνων ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως θα πρέπει η Κομισιό να θεωρήσει ότι το διάστημα αυτό, η προθεσμία αυτή είναι εύλογη προθεσμία. Αυτό θα το φροντίσουμε εμείς. Θα το ελέγξουμε δηλαδή. Επίσης θα πρέπει να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, που αφορούν ε, την χωματερή του Τερτσίνιο. Καταρχάς, ε, η οδηγία για, τις, για τους χιτά δεν απαγορεύει την λειτουργία χωματερών σε ένα εθνικό πάρκο και δεν το απαγορεύει ρητά. Όμως υπάρχει η οδηγία για habitat, για τους οικοτόπους, που προβλέπει ότι εφόσον ε, δημιουργούνται για λόγους... Ε, συμφέροντος της περιοχής ε, λοιπόν, εφόσον δημιουργείται τέτοιου είδους χωματερές σε ένα πάρκο ε, που ανήκει στο Natura 2000, θα πρέπει να ε, αξιολογηθούν οι εγκαταστάσεις αυτές με βάση το άρθρο 2.3 και 2.4 της οδηγίας. Όπως σας είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, όλα όσα θα γίνουν ε, από τις 4 Μαρτίου και μετά για να ε, εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση θα πρέπει να γίνει με κάθε σεβασμό της ε, κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Προφανώς εδώ μιλάμε για, για την επεξεργασία των αποβλήτων μένα, αλλά πρέπει να γίνουν σεβαστέ και οι διατάξεις των υπολείπων οδηγιών που αφορούν το περιβάλλον. Τώρα, να απαντήσω στον κύριο Ριβελίνη για τις κυρώσεις και τα πρόστιμα. Το δικαστήριο επιβάλλει τα πρόστιμα, η Κομισιό όταν παραπέμπει μία μια υπόθεση στην, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προτείνει κάποια πρόστιμα, όμως το δικαστήριο είναι ελεύθερο να αποφασίσει. Εφόσον οποιαδήποτε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απευθύνεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, είναι καθήκον του κράτους μέλους να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί τα πρόστιμα αυτά τα πρόσημα τα οποία του έχουν επιβληθεί. Πιστεύω ότι απήντησα στις διάφορες ερωτήσεις, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπουτσέλα. Τώρα, θα ήθελα να καλωσορίσω τους επισκέπτες σε δουλειά που έχουμε εδώ, που έχουν προσκληθεί από, τη, από το γραφείο μας στο Παρίσι. Θα ήθελα να τους καλωσορίσω εδώ. Αν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, υπάρχει ακόμα χρόνος για ερωτήσεις. Σαντρίν Μπελιέ έχει άλλη ερώτηση για την βιοπικιλότητα. Η Σαντρίν Μπελή όμως δεν είναι εδώ. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η κυρία Καρίν Κανερβάση ούτε και είναι εδώ όμως. Α. Ρίτσαρ Σίμπερ όμως. Είναι εδώ για την οδηγία πλαίσιο για τα υδάτα. Τρεις ερωτήσεις έχω εγώ για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν και να δημοσιεύουν σχέδια διαχείριση λεκάνη απορρή ποταμού. Η ερώτησή μου είναι ποια κράτη-μέλη έχουν ήδη δημοσιεύσει τα δικά του σχέδια διαχείριση λεκάνη απορρή ποταμού και πόσα σχέδια διαχείριση λεκάνη απορρή ποταμού έχουν δημοσιευθεί σήμερα και συνάδουν τα σχέδια με τι κατευθυντήριε γραμμέ τη οδική πλαισίου για τα ύδατα. Η άλλη ερώτηση έχει να κάνει με τον κανονισμό REACH. Μπορείτε σας παρακαλώ να σχολιάσετε ποια είναι η σημερινή κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη αναθεώρηση του κανονισμού και αν ναι, σε τι χρονικό πλαίσιο. Και τέλος θεωρεί η Επιτροπή ότι υπάρχει ανάγκη επέκταση του κανονισμού REACH. Η τελευταία ερώτηση του κ. Ζέμπερ είναι το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που εξετάζει τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες, ε, τη βιοπικιλότητα, το περιβάλλον, την υγεία και τους φυσικούς σπόρους και τα πόβλητα. Προχωράει η εφαρμογή του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον σύμφωνα με το πρόγραμμα. Και σε ποιο βαθμό έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του. Αυτές είναι οι ερωτήσεις και εγώ θα πρόσθετα και κάτι ακόμα. Επίτροπη, μίλησε για τη σύμβαση του και για τη συμμετοχή της κοινωνίας. Ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν. Η συμμετοχή της κοινωνίας ε, στις διαδικασίες αξιολόγησης ε, περιβάλλοντος είναι αποτελεσματική. Θεωρεί η Κομισιόν ότι πρόκειται για κάτι καθαρά τυπικό ή ότι πρόκειται για ένα πραγματικά αποτελεσματικό μέσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δυστυχώς δεν θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε σήμερα όλα τα σημεία αυτά. Θα πρέπει να περιμένουμε να το κάνουμε την επόμενη φορά. Αν μπορεί όμως η Επιτροπή να απαντήσει στο τρίτο ερώτημα. Γιούλιος Γκασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. τρία συγκεκριμένα ερωτήματα από τις οδηγίες πλαίσιο για τα ύδατα. Είναι το ποια κράτη-μέλη έχουν ήδη δημοσιεύσει εγκαίρω τα σχέδια διαχείριση λεκάνης απορροών ποταμών, πόσα σχέδια έχουν δημοσιευθεί και αν τα σχέδια συνάδουν με τι κατευθυντήριε γραμμέ τη οδηγία πλαισίου για τα ύδατα. Για την πρώτη ερώτηση, 12 κράτη-μέλη δημοσίευσαν εγκαίρως τα σχέδιά τους εντός της προθεσμίας ε, και έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2010. Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Γαλλία, Λετωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι χώρες που έχουν δημοσιεύσει λοιπόν εγκαίρως τα σχέδιά τους. Τέσσερα κράτη-μέλη έχουν ε, κοινοποιήσει τα σχέδιά τους, αλλά μετά την ε, προθεσμία, η Εσθονία, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Ιταλία. Και ξεκινήσαμε διαδικασίες επί παραβάση κατά των υπολείπων 11 κρατών μελών που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι για δύο υποθέσεις, την υπόθεση κατά του Βελγίου και της Λιθουανίας, μιλάμε για εν μέρη έλλειψη εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, γιατί τα δύο αυτά κράτη-μέλη έχουν υποβάλει κάποια σχέδια διαχείρισης, αλλά δεν καλύπτουν τα σχέδια αυτά όλη την επικράτεια των χωρών αυτών. Για τη δεύτερη ερώτηση, πόσα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού έχουν δημοσιευθεί σήμερα, πρέπει να πω ότι έχουμε λάβει 110 σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και μας λείπουν 66. Επιπλέον, έχουμε λάβει κάποιες κοινοποιήσεις για την έγκριση διεθνών σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Και για την τελευταία ερώτηση τώρα, για το κατά πόσο συνάδουν τα σχέδια με τις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Ήδη αρχίσαμε την αξιολόγηση του κατά πόσο τα σχέδια που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας, αλλά ακόμη πρέπει να συνεχίσουμε την εξέταση και έχουμε προβλέψει και διμερείς επαφές με τα κράτη-μέλη για το 2011. Και αν δούμε ότι κάποια από τα σχέδια δεν συνάδουν με την οδηγία, θα ξεκινήσουν διαδικασίες επί Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια έκθεση αξιολογώντας την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Και η έκθεση αυτή θα είναι τμήμα του σχεδίου του 2012 για την αδιάσωση των υδάτων στην Ευρώπη γενικότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής γιατί είσαστε και πάντοτε παρόν στην Επιτροπή μας και τα τελευταία 8 χρόνια, 8 χρόνια μας ε, απαντάτε στις ερωτήσεις μας ενώ τώρα θα πάτε σε νέα θέση. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στην καινούργια σας θέση και σας ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... πρέπει να πούμε ότι είναι μια συζήτηση που θα τη συνεχίσουμε και σε μελλοντικές συνεδριάσεις. Και πρέπει να πούμε τώρα πότε θα είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. 24 έως 26 Ιανουαρίου του 2011. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος της συνεδρίασης.